Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία. Έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Θα πάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 12. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας, υπεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού, Η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την οδηγία υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια στις 2 Απριλίου του 2009. Στην πρώτερη θητεία, στα πλαίσια διαδικασίας διαβούλευσης, με τη θέση ισχύ όμως της συνθήκης της τώρα έχουμε τη σύμφωνη γνώμη και ο κ. Ρωμέβα Ιρουέδα έχει καθοριστεί εισηγητής. Εκτιμούμε τα μάλα την προθυμία της Βελικής Προεδρίας να μας εξηγήσει την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου αυτού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις απόψεις της και μετά θα εξαχθεί σύντομη συζήτηση, αν μας επιτρέπει ο χρόνος, και μετά ο Διευθυντής της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, ο κ. Μόρτα Κυρίουγκ, θα μας παρουσιάσει τη νέα έκθεση του φορέα αυτού όσον αφορά τη διάκριση για λόγους ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, ισότητας των φύλων και λοιπά. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Ρωμέβα Ιρουέδα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εκ νέου το θέμα. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίας που δέχτηκε να ανταλλάξουμε απόψεις, όχι μόνο όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά και να προβληματιστούμε, να κάνουμε μια αποτίμηση του τι έχει γίνει και πού μπορούμε να πάμε. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι όπως αναφέρθηκε, έχουμε ήδη ένα κείμενο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία, στα πέσεις διαδικασίας διαβούλευσης και μέχρι τώρα οι ομάδες ε, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτό ως βάση της ε, θέσης μας. Τώρα βέβαια στο Συμβούλιο είναι το μπαλάκι και θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί. Το παρακολουθήσαμε το θέμα κατά διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και ελπίζουμε να έχουμε και καλές ειδήσει από τη Βελγική Προεδρία, όμως επικρατεί σε πολλούς από εμά το συνέστημα ότι είναι υπερβολικά αργή η πρόοδος και πολλοί από εμά βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Πολλές ομάδες βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Θέλαμε να κινηθούμε ταχύτερα. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό ενθαρρύνω όχι μόνο τα κράτη-μέλη μέσω του Συμβουλίου, αλλά και τους συναδέλφους, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και να συνεχιστεί η πρόοδος. Εξακολουθούν να απομένουν κάποια προβλήματα όσον αφορά το περιεχόμενο. Βασικά όμως υπάρχει και πίσω από αυτό ένα βασικό πολιτικό πρόβλημα, δεν είναι κάτι καινούριο. Το γνωρίζουμε από το παρελθόν και εμείς σαν πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο αναμένεται να βοηθήσουμε να βρεθεί μια λύση. Ας ακούσουμε πρώτα τι έχει να πει το Συμβούλιο και μετά με παρούσες διάφορες ομάδες μπορεί να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με το πώς το Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή μπορούμε να κινηθούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ας ακούσουμε την κυρία Περνό από την Βελγική Προεδρία. Καλημέρα σε όλους, θα μιλήσω Ολλανδικά. Καλημέρα, ευχαριστώ που μας καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες ε, της Βελγικής Προεδρίας ε, σε σχέση με αυτή την οδηγία. Αλλά πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση. Ξέρετε πως αυτή η οδηγία προβλέπει την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκείας πευθύσεων ηλικίας αναπηρίας και σεξουαλικού προσανατολισμού και είναι δύσκολη η οδηγία για διάφορους λόγους. Είναι δύσκολη για λόγους ουσίας, περιεχομένου, πολιτικούς, αλλά και για λόγους τεχνικούς. Και γιατί ε, σήμερα αντιμετωπίζουμε Συμβούλιο ένα αριθμό κρατών μελών που αυτή τη στιγμή από πολιτική σκοπιά δεν είναι σε θέση να στηρίξουν μια τέτοια οδηγία και να της δώσουν και προτεραιότητα. Και αυτή είναι μια κατάσταση η οποία μας λυπεί αλλά είναι η σημερινή πραγματικότητα. Ποιοι είναι τώρα οι λόγοι για αυτές τις επιφυλάξεις αυτών των κρατών μελών. και Έχουν τρεις ε, ειδικού ε, λόγους που αναφέρουν συνεχώς. Είναι η επικουρικότητα, η αναλογικότητα και η νομική ανασφάλεια. Για το τελευταίο ζήτημα υπάρχουν διαφοροί όροι που χρησιμοποιούνται και κυρίως βασίζονται σε αποφάσεις ε, του ΔΕΚ για να δώσουν κάποιες ερμηνείες ε, κάποιων λέξεων όρων στην ε, οδηγία που τους ανισχούν. Παραδείγματο χάρη για την κοινωνική ασφάλεια, εάν το δούμε αυτό μαζί με την ηλικία, αυτό που ανισχύει τα κράτη-μέλη, είναι πως το δικό του σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ε, αναφέρεται σε συγκεκριμένες ε, ηλικιακές κατηγορίες, κάτι το οποίο δεν θα είναι δυνατόν να γίνεται πλέον στο μέλλον. Εάν μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε κάποια... το να μπορέσουμε να έχουμε κάποια νομική ασφάλεια, είναι κάτι το οποίο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι σε πολιτικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα προβληματική αυτή η οδηγία στο Συμβούλιο και άρα λόγω της στάσεως τριών κρατών μελών δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα στο Συμβούλιο. Τι αποφάσισε λοιπόν να κάνει η Βελγική Προεδρία. Κοιτάξτε, επειδή είδαμε πως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε πολιτικό επίπεδο, στραφήκαμε στην τεχνική πλευρά για να επιτευχθεί εκεί κάποια πρόοδος. Τι κάναμε, βγάλαμε δύο θέματα από την οδηγία και προσπαθήσαμε με βάση αναλυτική έρευνα, αξιολόγηση και μια πιο θεματική ε, προσέγγιση να ασχοληθούμε με δύο θέματα. Και το ένα είναι οι οικονομικές υπηρεσίες, οι εξαιρέσεις δηλαδή που θα πρέπει να γίνουν με βάση ηλικία και αναπηρία στις ε, οικονομικές υπηρεσίες και το δεύτερο αντικείμενο είναι η στέγαση, η πρόσβαση στη στέγαση και τι ε, εννοούμε εδώ πέρα και ποιες, για ποιες συγκεκριμένες κατοικίες μιλάμε. Οπότε εργαστήκαμε περισσότερο στο τεχνικό επίπεδο με βάση την έρευνα και αυτό έγινε σε συνεργασία με μη κυβερνητικού οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα αναφέρω μία εδώ πέρα, την ε, ε, η LGB, την κοινωνική πλατφόρμα και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας. Και είχαμε συνεχείς ε, συνεδριάσεις στην ομάδα κοινωνικών υποθέσεων και συναντήσεις με τις ΜΚΟ έτσι ώστε να μας συμβουλεύσουν και προσπαθήσαμε έτσι να σημειώσουμε κάποια πρόοδο στο τεχνικό επίπεδο. Τώρα, Εάν δούμε τα συγκεκριμένα τεχνικά σημεία που είδαμε στις οικονομικές υπηρεσίες και τη στέγαση, ας δούμε τι κάναμε. Τι κάναμε πρώτα για τις οικονομικές υπηρεσίες. Ευτυχώς η Κομισιόν είχε παραγγείλει μια έρευνα στην οποία νομίζω θα επανέλθει για, σε μια συμβουλευτική εταιρεία η οποία είχε κάνει μια έρευνα ουδέτερη στα κράτη-μέλη για να δει σε ποιο βαθμό οι διάφορες διακρίσεις όπως η ηλικία, αναπηρία κτλ. χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ε, και τις ε, τράπεζες για να κάνουν εξαιρέσεις. Με βάση αυτή την έρευνα η Βελγική Προεδρία έστειλε ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη το είδαν αυτό πολύ ε, θετικά και έκαναν αρκετά καλή δουλειά. Δηλαδή έκαναν με βάση το ερωτηματολόγιο είδαν πώς ακριβώς δουλεύουν οι ασφαλιστικές εταιρείε και οι τράπεζες στα κράτη-μέλη. Και τι είδαμε μετά. Είδαμε πως ε, οι τραπεζικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν την αναπηρία ως μια δυνατότητα για να προσφέρουν μια εξαίρεση, για να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάκρισης δηλαδή και ε, μπορέσαμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη είναι πως περισσότερη σημασία έχει η κατάσταση της υγείας και όχι η ίδια η αναπηρία. Δεν σημαίνει πως ε, η αναπηρία σημαίνει κίνδυνο ή δυσκολία ε, παραδείγματο χάρη σε ένα δάνειο στεγαστικό ή μια ασφάλιση αυτοκινήτου. Και είπαμε, εάν, πρέπει, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εξαίρεση, αυτό πρέπει να γίνει με βάση δεδομένα ή αναλογιστικές αρχές. Και πρέπει να είναι βεβαίως αξιόπιστα τα δεδομένα και ακριβή και ελέγξιμα. Οπότε μετά προτείναμε ένα νέο ε, κείμενο, ειδικά όσον αφορά το άρθρο 2.7 και ξέρω πως εδώ η Κομισιόν έχει προτείνει μια αλλαγή. Κάτι το οποίο ήταν σημαντικό εντός των οικονομικών υπηρεσιών ήταν βεβαίως και η διαφάνεια. Διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή πως πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες δεν έχουν διαφάνεια όταν ε, αρνούνται να δώσουν ε, ένα δάνειο ή να ασφαλίσουν κάποιον. Θα πρέπει κάποιος να μπορεί να κάνει μια καταγγελία είτε σε κάποιο συνήγορο του καταναλωτή, είτε σε κάποιο σύνολο, σύνδεσμο καταναλωτών, για να μπορέσει να μάθει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ και είχαμε μια συγκεκριμένη πρόταση και προσθέσαμε στο άρθρο 2.7 ένα εκτιμώντας για να πούμε πως θα πρέπει όλοι να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ασφάλειες. Αυτό όσον αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες. Μετά έρχομαι στο θέμα της στέγασης. Εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε τι εννοούμε με τη στέγαση, γιατί υπάρχει και η ιδιωτική και η δημόσια και η κοινωνική στέγαση ε, είναι στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Και εδώ πέρα τα κράτη-μέλη εργάστηκαν με βάση ένα ερωτηματολόγιο και μπορώ να πω πως και εδώ πέρα είχαμε μια πολύ θετική απάντηση, αντίδραση από τα κράτη-μέλη και έκαναμε και εδώ πέρα μια νέα πρόταση διατύπωση με βάση αυτά τα οποία μας είπαν τα κράτη-μέλη και είπαμε πως κοιτάξτε ίσως είναι καλό να δοθεί μια εξαίρεση με βάση βεβαίως την προστασία της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής. Τι εννοούμε ακριβώς εδώ πέρα. Όταν κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας κατοικίας και εκεί πέρα ενοικιάζεται ένα δωμάτιο, τότε θα πρέπει βεβαίως να έχει κάποιο περιθώριο ο ιδιοκτήτης να αποφασίσει ποιον θα βάλει σπίτι του από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή θα πρέπει να αποτελέσουν ε, μία εξαίρεση ε, όσον αφορά την απαγόρευση διάκρισης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η κοινωνική ε, στέγη, η οποία επίσης θεωρούν πως θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εφαρμογής. Ούτως ή άλλως στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιας ή ιδιωτικής ή κοινωνικής στέγασης, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη και η κοινωνική στέγαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Γιατί αποτελεί μέρος κοινωνικής προστασίας. Και, κάτι τελευταίο, η πρόσβαση στην ε, στέγαση και η μια ε, λογική προσαρμογή την οποία μπορεί να ζητήσει ένας ανάπηρος αλλά ε, το θέμα είναι ως ποιο βαθμό μπορούμε να αναγκάσουμε τον ιδιοκτήτη μιας κατοικίας να κάνει τέτοιες προσαρμογές στην κατοικία για έναν ανάπηρο. Και εκεί πέρα τεχνικά μπήκαμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας και είδαμε την ισορροπία που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ αφενός του αναπήρου ατόμου και αφετέρου την ε, ελευθερία του ιδιοκτήτη και εκεί πέρα κάναμε κάποιες προτάσεις κειμένου ακριβώς για να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Αυτά είναι δύο μεγάλα θέματα που απασχόλησαν την ε, Προεδρία μας. Όπως σας είπαμε, βάση έρευνα, ερωτηματολόγια και είχε θετικό αποτέλεσμα υπό την έννοια πως μπορούσαμε να εργαστούμε εις βάθος, πως τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν μια θετική στάση και δεν ε, άρχισαν να υπερασπίζουν κάποιες θέσεις αλλά συζήτησαν ανοιχτά. Και ελπίζουμε η Ουγγρική Προεδρία να ακολουθήσει αυτό τον τρόπο εργασίας έτσι ώστε εάν μπορούμε μία μέρα πολιτικά να προχωρήσουμε παραπέρα να είναι τεχνικά ήδη πιο προχωρημένη η οδηγία να επισημάνω στα μέλη της Επιτροπής σας πως εκτός από αυτή την οδηγία η Βελγική Προεδρία οργάνωσε και τη Σύνοδο Κορυφής Ισότητας με 500 εκπροσώπους από όλες τις ΜΚΟ και τα κρατημέλη. Μια σημαντική δραστηριότητα, κάναμε και μια αξιολόγηση των δύο οδηγιών που αφορούν την μη διακριτική μεταχείριση στο χώρο εργασίας για να χρησιμεύσει αυτό ως υπόδειγμα ε, για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά μια τέτοια οδηγία και να έχουμε μια θετική εξέλιξη όταν θα εγκριθεί. ελπίζω να σας ενημέρωσα λοιπόν επαρκώς και αν θέλετε κάποια ερώτηση είμαι στη διάθεσή σα. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος του κύριο Όλσον από την Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, ξέρω ότι η Μέσια διάταξη σας είναι φορτωμένη. Η Κομισιόν επιβεβαιώνει 100% τα όσα ανέφερε η Βελική Προεδρία. Ευχαριστούμε την Βελική Προεδρία για την προσέγγιση που διάλεξε. Έχει αφιερώσει χρόνο, έχει αφιερώσει προσωπικό. Είναι δύσκολο να γίνει πρόοδος ε, μέσα σε μία προεδρία ε, για οποιοδήποτε δύσκολο θέμα. Ευχαριστούμε λοιπόν την Βελική Προεδρία. Να προσθέσω ότι εκτός των τεχνικών συζητήσεων η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κυρία Ρέντινγκ έχει αφιερώσει πολλή προσπάθεια σε υψηλό επίπεδο συναντήσεις με υπουργούς και με αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων ορισμένων από τις πιο σημαντικές για αυτό το ζήτημα χώρες για να αναζητηθούν λύσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν βρεθεί. Δεν έχει επιτευχθεί δηλαδή πολιτική πρόοδο. Συνεπώς συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και να διευκρινίσουμε σε, πολιτικό, σε τεχνικό επίπεδο, συγγνώμη, αναμένοντας ε, πρόοδο και στο πολιτικό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι στις επόμενες προεδρίες, Ουγγρική και Πολωνική, θα συνεχιστεί η προσπάθεια και στα δύο αυτά επίπεδα. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική ερώτηση υπάρχει. Ευχαριστώ. Ωραία. Οι συνάλφοι θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Κύριος Ντεγιόν. Και βέβαια ο εισηγητής ο κύριος Ρωμέβα. Κυρία Ίνφελτ. Και μετά ξανά στον εισηγητή. Ο κύριος Ντεγιόν καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήξερα πως δεν υπάρχει πρόοδος στο Συμβούλιο, αλλά είναι απογοητευτικό να ξανακούμε το ίδιο πράγμα. Έχουμε βεβαίως και την υπόθεση του, της υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έκανε μια καλή προσπάθεια η Βελγική Προεδρία, αλλά θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν ε, και η Βελική Προεδρία αν είναι ε, αισιόδοξε για τις επόμενες προεδρίες και αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα οποία στηρίζονται και δεύτερον η εξαίρεση στην στέγαση για λόγους ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής κάτι το οποίο ε, δεν βρίσκω τόσο θετικό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη και αυτό σημαίνει πως ε, εάν κάποιος ξέρω εγώ, έχει προκατάληψη έναντι των μαύρων ή των Εβραίων ή δεν ξέρω εγώ ποιανού ή άλλες μειονότητες μπορεί να πει όχι δεν σου νοικιάζω το δωμάτιο. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν πού φτάνει αυτή η οδηγία γιατί δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να αποτελέσει κάτι τέτοιο δικαιολογία τη στιγμή που ε, δηλαδή θα, θα βάλεις κάποιο ξένο στο σπίτι σου έναντι χρημάτων να βάζεις ε, τέτοιους ε, όρους. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διάκριση. Μπορείς άμα δεν θες να μην νοικιάσεις το δωμάτιο. Θα ήθελα λοιπόν μια διευκρίνηση εδώ πέρα γιατί μου φαίνεται λίγο επικίνδυνο αυτό. Και τέλος, θεωρεί η Βελγική Προεδρία πως ε, είναι ευκολότερο παραδείγματος χάρη να προχωρήσουμε όσον αφορά την αναπηρία σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό όσον αφορά τα άλλα κράτη-μέλη. Πώς έχει ακριβώς η κατάσταση. Ευχαριστώ. The next question, Mrs. Κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ας μιλήσω και εγώ Ολλανδικά. Ευχαριστούμε την Βελγική Προεδρία που με ρεαλιστικό τρόπο είδε αυτό το θέμα που τελικά είναι μια δύνατη αποστολή. Είναι λογικό να προσπαθεί να κάνει βήμα-βήμα πρόοδο στα τεχνικά ζητήματα, αλλά βεβαίως ξέρουμε πως αυτή η προσέγγιση έχει όρια, γιατί τα προβλήματα δεν τεχνικά είναι πολιτικά. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. το συγκρίνουμε παραδείγματο χάρη με την Ευρωζώνη όπου λέμε όλοι ότι κάτι θέλουμε, θέλουμε ένα ταμείο διάσωσης, πρέπει να αλλάξει η συνθήκη, κανένα πρόβλημα θα το κάνουμε. Αλλά δεν γίνεται το ίδιο όταν μιλάμε για την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις τεχνικές λεπτομέρειες. Έτσι αυτό να το αναφέρω παρενθετικά ότι ε, να μας λένε μετά δηλαδή και οι τράπεζες ε, πως είναι επικίνδυνο να δανείζουν ε, σε ανάπηρους μετά από όλη αυτή την κρίση ε, εντάξει δεν είναι αυτός ο κίνδυνος που έχουν επομιστεί οι τράπεζες έτσι να το πω και λίγο κοινικά το Βέλγιο έχει νομίζω αρκετά καλό ιστορικό στο θέμα της προστασίας από τις διακρίσεις και από την αρχή όλης αυτής της διαδικασίας Αναρωτιέμαι αν θέλουμε πράγματι βεβαίως μια τέτοια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων και ταυτόχρονα Το θέμα είναι πως ε, τι θα κάνουμε με τις ε, πρακτικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και αν θα τις αντικαταστήσουμε και φοβάμαι πως ο κίνδυνος αυτός υπάρχει δηλαδή θα υπάρξει μείωση των ήδη υφισταμένων ε, ευεργετικών διατάξεων. δεν ξέρω αν σε άλλες περιπτώσεις θα εδραιωθούν οι πρακτικές των κυβερνήσεων οι οποίες δεν είναι τόσο λογικές. Ε, Ο εισηγητής. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βελική Προεδρία που ήταν παρούσα. Έχω παρακολουθήσει και τις δύο τελευταίες προεδρίες, την Ισπανική και τη Βελική, από πολύ κοντά. Και οι δύο έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία για να προχωρήσουμε και από ό,τι φαίνεται ε, υπάρχει εκ μέρου ορισμένων κυβερνήσεων ε, μια έλλειψη βούλησης και ε, μια, γίνεται μια προσπάθεια παρεμπόδισης πρόοδου. Αυτό είναι δυσάρεστο. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε κάτι, κάποιο θέμα σχετικό με την ουσία. ξέρω ότι δεν είναι πολιτικός ορθό να το λέμε, αλλά θα ήθελα να το πω θα πρέπει να βάλουμε, να δώσουμε όνομα, ονοματεπώνυμο για την ακρίβεια σε αυτούς που αντιδρούν. Διότι έχει σημασία να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι χώρες που αντιδρούν και για ποιο λόγο βέβαια δεν είναι υπέρ της πρόοδου αυτής της ε, οδηγίας. Ε, είναι απαραίτητη αυτή η διαφάνεια. Ξέρω ότι το Συμβούλιο δυσκολεύεται αν όχι ε, αδυνατή να ε, αποκαλύψει τέτοιου είδου στοιχεία. Ε, ξέρουμε βέβαια ε, ότι υπάρχει η Γερμανία, είναι το κράτο το οποίο γνωρίζουμε ότι αντιδρά. Θα θέλαμε να δούμε και ποια είναι τα υπόλοιπα. Δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέξω είναι το εξή. Ορισμένα από αυτά τα επιχειρήματα τα οποία υποτίθεται ότι προβάλλει το Συμβούλιο για να μην προχωρήσει το θέμα, έρχονται σε αντίθεση με την εθνική νομοθεσία πολλών από αυτέ τι χώρε. Για παράδειγμα, στην περίπτωση τη Γερμανίας. Η Γερμανία αντιδρά με μια ευρωπαϊκή οδηγία που διευρύνει δικαιώματα τα οποία ήδη υπάρχουν στη Γερμανία. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε γιατί, α, όπως έλεγε η Σοφή, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το να μην δεχόμαστε ως ευρωπαϊκό δικαίωμα την ισότητα στη μεταχείριση όταν αυτό το δικαίωμα ήδη υπάρχει στην ομοθεσία πολλών κρατών μελών. Συνεπώς δεν θα πρέπει τα δέντρα να μας εμποδίζουν να δούμε όλο το δάσος. Να μιλάμε δηλαδή για τα τεχνικά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα ουσίας είναι το δάσος. Επόμενη σκέψη είναι εξής. Το νέο νομικό πλαίσιο μας δίνει περισσότερα νομικά εργαλεία. Για παράδειγμα, η Σύμβαση του ορισμένου Εθνών για την Αναπηρία είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα, μπορούμε, θα μπορούσαμε να εργαστούμε, για παράδειγμα να σκεφτούμε πώς ε, θέλουμε να γίνουμε μέρος αυτής της σύμβασης. Πέμπτη ιδέα είναι εξή. Έχει λεχθεί επανειλημμένως και είναι αλήθεια ότι ε, τίθεται θέμα αναλογικότητας, ε, νομικής ασφάλειας και επικουρικότητας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν ορισμένες από αυτές τις ενδεχόμενες ε, αντιφάσεις έφτασαν στα δικαστήρια, Ελάχιστες ήταν οι δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν. Κάτι που δεν δικαιολογεί το επιχείρημα ότι υπάρχει κίνδυνος αναλογικότητας, επικορικότητας κλπ. Γιατί πολύ συχνά χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα, αλλά στην πράξη δεν έχει αποδειχθεί ότι ε, το σύστημα είναι περίπλοκο ή ότι πραγματικά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος που δεν μπορεί να αποφευθεί. Τελευταία σκέψη πολύ συχνά έχει χρησιμοποιηθεί ένα επιχείρημα το οποίο δεν το ακούσαμε σήμερα, αλλά το ακούμε. Το θέμα της οικονομικής κρίσης και του κόστους που θα συνεπάγει η εφαρμογή αυτής της οδηγίας, ε, ιδιαίτερα ορισμένες πτυχές της, όπως η πρόσβαση στην στέγη και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι Η τελευταία εκδοχή του κειμένου αλλά και άλλες προηγούμενες ε, δίνει και οι προηγούμενες επίσης έδιναν ε, μεγάλα χρονικά περιθώρια στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Παλιότερα και το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο είχαν δεχτεί προθεσμίες εφαρμογής ε, πολύ μακρινές. Συνεπώς ούτε αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο, ε, ε, επιχείρημα το κόστος. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν στο Συμβούλιο να το χρησιμοποιούν, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση αυτού του επιχειρήματος, διότι στην πράξη το ερώτημα είναι αν δεχτούμε ότι η μη διάκριση έχει ένα κόστος, μην ξεχνάμε ότι έχει κόστος και θα πρέπει να το συγκρίνουμε και ατομικό και οικονομικό κόστος η εφαρμογή διακρίσεων. Αυτά θα πρέπει λοιπόν να τα έχουμε υπόψη μας για να έχουμε στο μυαλό μας όλο το πανόραμα. Ασφαλώς και υπάρχουν τεχνικά θέματα, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πρόσβαση στη στέγη. Χαίρομαι που ακούω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αν είχα καταλάβει καλά κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας αλλά ενδεχομένω και της Βελικής Προεδρίας. Οπότε, δημιουργεί οπότε παρουσιαζόταν μία δυσκολία στην επόμενη συνεδρίαση οι λύσεις προτείνονταν δημιουργούσαν πολύ περισσότερα προβλήματα αλλά χαίρομαι που ε, προχωρήσαμε σε τεχνικό επίπεδο αυτό το εξάμεινο. Επιμένω ότι ε, για αυτό το θέμα η, η βούληση της Επιτροπής μας και νομίζω, θέλω να πιστεύω και του Κοινοβουλίου υπάρχει, πρέπει να προχωρήσουμε και πιστεύω λίγο πιο γρήγορα. Γιατί, γιατί το αίτημα έρχεται από την κοινωνία, γιατί εδώ και πολύ καιρό τα θύματα αυτών των διακρίσεων το ζητούν και γιατί, επιτρέψτε μου να το πω, το θέμα αυτό θα βελτιώσει την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εποχή που αυτή η αξιοπιστία αφισβητείται. Τελειώνω με ένα αίτημα και προς την, προς Προεδρία του Συμβουλίου. Θα ήθελα τέτοιου είδου συναντήσεις ενημερωτικές για το στάδιο των Ανασιών να γίνονται πιο τακτικά, τουλάχιστον μία φορά δυνατόν κάθε εξάμεινο με την κάθε διαφορετική προεδρία. Παρακαλώ το θέμα αυτό να μην εξαφανιστεί από την μερίσια διάταξη επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο θέλει να πει κάτι. Ναι, θα αναφερθώ σε κάποια ερωτήματα και δεν ξέρω μετά αν θέλω να απαντήσει η Κομισιόν. Ο κύριος Ντεγιόγκ ρώτησε ειδικά για τους Ούγγρους τι θα κάνουν με το θέμα αυτό. Ξέρετε πως στην Ουγγαρία μόλις ανέλαβε η κυβέρνηση καθήκοντα και δεν έχουν καθοριστεί οι αρμοδιότητες των Υπουργείων. Από τους Ούγγρους συναδέλφους μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για το πρόγραμμά τους. Οπότε είναι δύσκολο να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί οι ίδιοι οι Ούγγροι το συζητάνε εσωτερικά ακόμα για το ποιος ακριβώς θα είναι ο αρμόδιος Κατόπιν για την εξαίρεση αυτή που θα δοθεί για την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή να σας πω έπρεπε ίσως να διευκρινίσω. Δεν είναι το θέμα πως κάθε ιδιωτική, αν θέλετε, οικογενειακή ζωή θα αποτελέσει εξαίρεση. Όταν μιλάμε για την στέγαση, όταν ε, μιλάμε για ένα σπίτι με κοινή κουζίνα, κοινό μπάνιο, ε, και όπου όντως δηλαδή μιλάμε για ιδιωτική ζωή και για αυτή την περίπτωση θα μπορέσουμε να δώσουμε μια περιορισμένη εξαίρεση, αλλά από τη στιγμή την οποία κάποιος νικιάζει το διαμέρισμά του, έστω και αν αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ε, κατοικίας ε, μέσω ενός πρακτορείου, τότε βεβαίω μιλάμε για κάτι το οποίο είναι στη δημόσια σφαίρα και ισχύουν όλα αυτά. Οπότε μιλάμε για πολύ περιορισμένη εξαίρεση. Εκεί τώρα όπου κάποιο κράτος μέλος είναι πιο ευαίσθητο για μια εξαίρεση, κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη σεξουαλική... Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι τόσο σημαντικός ή είναι πιο σημαντική αναπηρία. Αλλά δεν έχουμε την αίσθηση πως ε, κάνουν κάποια διάκριση τα κράτη-μέλη όσον αφορά το είδος της ε, διακρίσεις που γίνεται. Απλά αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ είναι πως ε, πράγματι ορισμένα πράγματα λαμβάνουν περισσότερη προσοχή. Τέλος, για τον ε, κίνδυνο να περιοριστούν καλές πρακτικές και να μείνουν μόνο οι κακές πρακτικές. Κοιτάξτε, Ακριβώς αυτό το οποίο προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε είναι να περιοριστούν οι λανθασμένες αυτές τις πρακτικές και ε, να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια έτσι ώστε όταν υπάρχει μια απόκληση η οποία θα επιτρέπεται να είναι περιορισμένη, να ξέρουμε γιατί ισχύει, να μπορούν να αποδειχθούν οι λόγοι μέσω αξιόπιστων δεδομένων κτλ. Και άρα μεγαλύτερη διαφάνεια. Δηλαδή για τις λανθασμένες πρακτικές ακριβώς αντιμετωπίζουμε. Για τις υφιστάμενες πρακτικές ε, σε κάποιες τράπεζες και ε, ασφαλιστικές εταιρείε πρέπει να τις περιορίσουμε και βεβαίως να τις δικαιολογήσουν για να είναι προφανές το τι συμβαίνει για όλους και να υπάρχει μια διαφάνεια στην πολιτική των ασφαλιστικών ε, εταιριών. Ελπίζω να σας διαφώτισα. Uh, Ευχαριστώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει να δώσει κάποια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα και πάλι όσον αφορά το θέμα των εξαιρέσεων και τη συγκεκριμένη εξαίρεση που έθιξε ο κ. Γιόγκ, έχω να πω το εξή. οι πρώτες Ευρωπαϊκής και η πλήρης γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου λαμβάνουν υπόψη ότι έχουμε χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρέπει να φροντίσουμε η πρόταση να σέβεται τη χάρτα. Και το δικαίωμα της προστασίας ιδιωτικής ζωής είναι ένα ζήτημα. Όπως είπε και η Προεδρία, πρέπει να αντικατοπτρίζονται διάφορα θεμελιώδη δικαιώματα και η ισορροπία της προτάσεως πιστεύω ότι είναι ορθή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να αποδυναμώσει το κείμενο και να καταλήξουμε σε κάτι που δεν θα εμπεριέχει ισορροπία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όσον αφορά τους διάφορους λόγους, εμείς πιστεύουμε ακραδάτο ότι αυτή η πρόταση πρέπει να παραμείνει ενιαία. Να μην προβάλλουμε ένα επιχείρημα έναντι άλλου για θέματα ασφαλείας δικαίου, για τα οποία φροντίζει πάντα το Συμβούλιο, για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων, πρέπει η οδηγία να παραμείνει ενιαία. Δεν πρέπει να υπάρξει νέα ιεράρχηση. Και τώρα, αν κάποια ζητήματα δυσκολότερα από άλλα, τα θέματα του ορίου ηλικίας Φερρυπίν είναι κάτι που υπάρχει. Και εκτός της αγοράς εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση Φερρυπίν. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί όταν θα συζητήσουμε το τελικό κείμενο τη οδηγία, Έχουμε και το θέμα της προσβασιμότητας. Ανέφερε και ο Ρωμέβα τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων με αναπηρίες. Και θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το θέμα της προσβασιμότητας θα συμπεριληφθεί. Είναι δαπανηρό, χρειάζεται ίσως και μακρότερη περίοδος προσαρμογής και εφαρμογής. Αλλά το σημαντικότερο είναι να παραμείνει ένα ενίο σύνολο η οδηγία. Ευχαριστώ κύριε Όλσον. Η Σόφι Ιντβέλτ, αλλά πάρα πολύ σύντομα, Σόφι. Ναι, Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα. Να ξεκαθαρίσω προς τη Βελική Προεδρία κάτι. Δεν αναφερόμουν σε εξαιρέσει από επιχειρήσει ασφαλιστικέ εταιρείε και τράπεζε. Αναφερόμουν στι εξαιρέσει που τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αποσπάσουν για το μίσο που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό με ανησυχεί. Καλώς λέει Πρόεδρος. Στον κύριο Κύρα μου θα δώσω το λόγο τον πρόεδρο της Υπηρεσίας τα Θεμελιώδη Δικαιώματα για να κάνει μια παρουσίαση της εκθέσεως του φορέα αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι έχουμε χρονικά όρια στενά, οπότε θα αναφέρω κάποια βασικά στοιχεία. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ και να παρουσιάσω την νέα μας έκθεση σχετικά με την ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, ανεξάρτητα ε, από ομοφοβία, τρανσφοβία και, και σεξουαλικό προσανατολισμό. Είναι η πρώτη έκθεση που ετοίμασε η υπηρεσία μας. Αναλύει τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν επί νομικής βάσης. Θα κάνουμε στο μέλλον πολύ περισσότερες εκθέσεις επί διαφόρων τομέων. Όταν εκπονούμε μια έκθεση, πολύ συχνά αποτελεί μια φωτογραφία του νομικού καθεστώτος ποια είναι η κοινωνιολογική επιτόπου κατάσταση. Και είναι ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. Μας δείχνει ποια είναι η κατάσταση. Προστιθέμενη αξία πετυχαίνουμε όταν εντοπίζουμε τάσεις. Όταν εσείς μπορείτε να δείτε ότι οι παρεμβάσεις σας ελπίζουμε ότι έχουν αποτελέσματα όσον αφορά την επιτόπου κατάσταση. Ή που δεν δεν έχουν κάποια αποτελέσματα οι παρεμβάσεις. Τι πηγαίνει καλά, τι δεν πηγαίνει καλά. Αυτή είναι η πρώτη έκθεση αυτού του είδους και εν συντομία θα πω ότι η έκθεση ε, περιέχει διάφορους τομείς που περιγράφονται και βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, βελτιώνονται, βελτιώνεται η νομοθεσία και καταργούνται διάφορα παλιά φαινόμενα, εξαλείφονται. Η πρώτη έκθεση ξεκίνησε το 2008 στην Επιτροπή σας. Τα στοιχεία χρονολογούνται το 2007 και τα στοιχεία που παρουσιάζουμε σήμερα φτάνουν μέχρι το καλοκαίρι του 2010. Αυτό είναι το χρονικό φάσμα που καλύπτουμε δύο με τρία χρόνια. Πρέπει να πηδήξω σε άλλο σημείο τώρα της παρουσίασής μου. η συνεχιζόμενη βία και η ποινικοποίηση των ατόμων αυτών που εξετάζουμε ε, είναι θέμα κυρίως όσον αφορά ε, τους διάφορους αμφιφιλόφιλους κατά τον τρανσέξουαλ και έχουμε επιδίνωση σε σχέση με την ε, προηγούμενη έκθεσή μας. 11 κράτη-μέλη θεωρούν ότι ε, η ομοφοβία είναι κάτι επιβαρυντικό στοιχείο σε, σε διάφορες υποθέσεις. Προσετέθησαν και δύο χώρες στον κατάλογο. Κάτι πιο θετικό, η Σκοτία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει συγκεκριμένους νόμους για τους τρανσέξουαλ στο ποινικό της δίκαιο. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η εφαρμογή της αρχής της ισότιμης αντιμετώπισης στα κράτη-μέλη. Θετικές εξελίξεις έχουμε όσον αφορά το θέμα αυτό. Βλέπουμε ποια είναι η τάση. 18 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαγορεύουν τη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε τομείς πέρα από την απασχόληση, όπως σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως ήδη συζητήσατε. Από 16 που είχαμε πριν από 3 χρόνια έχουμε 18 χώρες τώρα. Και 20 κράτη-μέλη, πριν είχαμε 18, άρα συν 2, οι εθνικοί φορείς την ισότητα που δημιουργήθηκαν βάσει της οδηγίας για την ισότητα καλύπτει και το σεξουαλικό προσανατολισμό και διάκριση εξαιτία αυτού. άλλη εξέλιξη στον την ισότιμη αντιμετώπιση, όσον αφορά την επανένωση οικογενειών και την ελεύθερη διακίνηση, είναι ότι τρία κράτη-μέλη τώρα, ρητά, τώρα κινούμεθα σε αντίθετη κατεύθυνση, τροποποίησαν την νομοθεσία τους και καθορίζουν ρητά ότι ο γάμος αφορά αποκλειστικά άτομα του αντιθέτου φίλου και μόνο. Και πολλά άλλα κράτη-μέλη αρνούνται την αναγνώριση ε, γάμου ομοφιλοφίλων ε, και που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που καλύπτει αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν μπορούν να απολαύσουν πλήρως το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και επανένωσης με εκείνους που αγαπούν στο νέο κράτος μέλος διαμονής, ανεξάρτητα από τον ε, γενετήσιο προσανατολισμό. Έχουμε λοιπόν αυτές τις χώρες που θεώρησαν αναγκαίο να ετοιμάσουν ειδική νομοθεσία όσον αυτό το θέμα. Διότι θα έλεγα ότι η γενική τάση που εντοπίζουμε είναι μια προοδευτική προσέγγιση. Τέσσερις νέες χώρες μετά το 2007 θέσπισαν νομοθεσία όσον αφορά το γάμο ομοφιλοφίλων και τρεις χώρες θέσπισαν νομοθεσία όσον αφορά τις επίσημα αναγνωρισμένες ε, συμβιώσεις. Οι τάση είναι προδευτική. Αναγνωρίζει γάμους ομοφιλοφίλων άμεσα ή τουλάχιστον επίσημη συμβίωση. Τρεις χώρες όμως κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση και με πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τρόπο. Πολλές από τις αρνητικές εξελίξεις που ανέφερα κροθυγός πάνε μαζί με τις θετικές εξελίξεις. Οι αρνητικές τάσεις απορρέουν από την ε, μονή που υπάρχει όσον αφορά την μυσαλλοδοξία και θα το εξετάσουμε αυτό στην επόμενη ε, ενημέρωσή μας όσον αφορά την κοινωνιολογική ε, έκθεση. Αυτό είναι το νομικό καθώς περιγράφουμε εδώ και θα δούμε τι αντιστοιχήση υπάρχει αυτών των φαινομένων στην κοινωνιολογική ανάλυση. Σε αυτή τη φάση συμπεραίνουμε ότι ότι υπάρχουν πολύ βαθιές ομοφοβικές τάσεις ε, σε κράτη-μέλη. Από τις έρευνές μας ε, βλέπουμε τι γίνεται και στην παιδεία. Ο τομέας της παιδείας, κυρίως ε, δημοτικό, δευτεροβάθμια παιδεία, εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντική τομής. Τελείωσε ο χρόνος μου, θα έλεγα πολλά περισσότερα. Διαβάστε όμως σας παρακαλώ την έκθεση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, πολλά διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις που βλέπετε τις εξελίξεις συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβάλλει στις περαιτέρω εξελίξεις και να δώσει όθηση στη νέα οριζόντια οδηγία που απαιτείται. Στα κράτη-μέλη είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η ιεράρχηση με βάση τη διάκριση αυτή. Και ελπίζω ότι οι επόμενες προεδρίες θα μπορέσουν να απαλλαγούν από αυτές τις διαφορές και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ κύριε Κύριο. Ευχαριστούμε που αφιερώσατε αυτό το χρόνο και ζητώ συγγνώμη που σας πιέσαμε χρονικά. Η κυρία Ιντβελτ θέλει να προσθέσει κάτι. Δεν θέλω να ξαναρχίσουμε συζήτηση. Η κυρία Ιντβελτ όμως θέλει να πει δύο λόγια. Δεν έχουμε χρόνο πολύ. Αν όμως έχετε να πείτε κάτι. Κυρία Μποσκούρτ. Έχω μπερδευτεί τώρα. Μπορούμε να, να θέσουμε ερωτήσεις. Τι γίνεται. Κάντε μία ερώτηση, αλλά δεν θα κάνουμε συζήτηση γιατί ο χρόνος τελειώνει. Ε, κρίμα, κρίμα. Μια που είναι εδώ ο κύριος Κέρομ που ήρθε να μας πει αυτά τα πράγματα και δεν μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του μετά για τον χρόνο. Ε, εν πάση περιπτώσει, δύο σύντομες ερωτήσεις. Τι γίνεται με τις υποψήφιες χώρες μιλήσει. Εσείς βεβαίως ασχολείστε με τις 27, αλλά οι υποψήφιες χώρες θέλουν να γίνουν μέλη. Και πρέπει να εκπληρώνουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερο ερώτημα. Ε, λέτε πως κάποια κράτη-μέλη ε, θεώρησαν την ομοφοβία ε, επιβαρυντικό παράγοντα στην ομοθεσία. τι γίνεται με την καταγραφή των εγκλημάτων ε, μίσους ε, κατά τη μέλη. Το είδατε αυτό και ποια είναι τα, τα συμπεράσματά σας. Ε, ε, έτσι κι αλλιώς θα φάμε μαζί με τον κύριο Κέρουμ, οπότε δεν υπάρχει θέμα, λέει η κυρία Αντφέλτ. Κύριος Δεγιόγκ. Uh, θα είμαι σύντομος, πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εδώ τον κύριο Κέρομ. Πραγματικά αξίζει επένους για αυτή του την έκθεση, για αυτή τους την έκθεση. Κατά τη διάρκεια του γεύματο θα συζητήσουμε πιο λεπτομερώ, αλλά να πω και το εξή. Στην Ολομέλεια έγινε μια συζήτηση με την Επιτροπό Ρέντινγκ την οποία μάλιστα ξεκίνησα εγώ, για το ζήτημα ότι ορισμένα κράτη-μέλη φαίνεται ότι αποκλείουν τους γάμους ε, ατόμων δύο φίλου από την εθνική του νομοθεσία. Και τότε σε εκείνη τη συζήτηση στην Ολομέλεια η Επίτροπος ε, Ρέντινγκ φάνηκε ε, να πιστεύει ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της οδηγίας ελεύθερης διακίνησης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κερμάν αν πιστεύει ότι αυτό είναι σωστό. Ακόμα περιμένουμε την απάντηση της Κομισιόν σε μια επιστολή που, μέσω της οποίας ε, τη ρωτούσαμε αν θα αναλάβει δράση εναντίον των κρατών μελών που εφαρμόζουν τέτοιου είδους περιορισμούς. Κύριο Κέρομα έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Για το θέμα των ε, υποψηφίων χωρών. Μέχρι στιγμής δεν κάνουμε δικές μας έρευνες στις υποψήφιες χώρες, αλλά το καλοκαίρι η Κροατία είναι παρατηρητής στην υπηρεσία μας, οπότε μπορούμε να κάνουμε τις ερευνές μας και στην Οκρατία, ελπίζουμε και στην πούγουδομου του χρόνου, η Τουρκία εκρεμεί και ίσως κάποια στιγμή αργότερα. Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον με την Κροατία θα κάνουμε αυτές τις έρευνες στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα, αλλά συμφωνώ μαζί σας, είναι σημαντικό να το δούμε, να δούμε και αυτές τις χώρες. Για την καταγραφή, τα, το, τα οποία είπατε για το, το επιβαρυντικό στοιχείο, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε γενικώ ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε με διάφορους τρόπους που αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τη συλλογή δεδομένων. για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα ζητήματα. Θα ήθελα να το δούμε αργότερα, αν γίνεται, για την ελευθερία διακίνησης και την επανένεση οικογενειών. Και στην προηγούμενη έκθεση και σε αυτήν θίξαμε το θέμα αυτό με βάση την οδηγία της ε, ελεύθερης ε, διακίνησης, αλλά θα αφήσω στην Κομισιόν την νομική ανάλυση και θα αναμείνω την ε, απάντησή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε κύριο. τώρα. Τελειώνουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και πριν περάσουμε στο σημείο 13 θα ήθελα να σας πω πως θέλω να εγκρίνετε την απόφαση των συντονιστών για τους εξής ε, εισηγητές. Η κυρία Χάουτα αλλά για την εφαρμογή του 1014 01 για την πρόσβαση στα έγγραφα. Ο κύριος Μπούζουτιλ για την απαλλαγή του προπολογισμού για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίε και τις Κομισιόν. Και την κυρία Ενιτφέλντ για τη συμφωνία με τον Καναδά για την χρήση δεδομένων αεροπορικών επιβατών. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, θέσπιση του Eurodac για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων αναδιατύπωση. Είναι φάκελος του πακέτου του ασύλου και τα επόμενα λεπτά θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης της πρότασης κανονισμού Eurodac που παρουσίασε 11 Οκτωβρίου 2010 η Κομισιόν η κυρία Μόνικα Μακοβέη είναι η συγγήτρια. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακοβέη να μας ερουσιάσει σχέδιο έκθεσης και μετά θα γίνει συζήτηση. Thank Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε η Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση για τον κανονισμό Eurodac στις 11 Οκτωβρίου του 2010 είναι η τρίτη πρόταση που αφορά αυτό το κείμενο μετά το Δεκέμβριο 2008 και το Σεπτέμβριο 2009 και σχετικέ σχετικές προτάσεις. Αυτή η πρόταση υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2010. Αφαιρεί την επιλογή χρήσεω για τις δυνάμει του νόμου που περιλαμβανόταν στην πρόταση του Σεπτεμβρίου του 2009, λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2009 και τις πρώτερες συζητήσεις του Συμβουλίου εισάγει δύο στοιχεία συμπροματικά. Στο άρθρο 18, παράγραφος 4, εισάγει την ανάγκη για έλεγχο των αυτομάτων αποτελεσμάτων α, θερμικών απεικονίσεων από ειδικό για τα ε, ε, αποτυπώματα και στο 24.1 υπάρχουν διάφορες διατάξεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή της Σύμβαση του Δουλίνου να συμπεριλαμβάνει στο φυλάδιο πληροφορίε δεχτυλικά αποτυπώματα. Το φυλάδιο που θα ετοιμαστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 τη Συμβάσεω του Δουβλίνου. Στο σχέδιο εκθέσεω που απεστάλει σε εσά την περασμένη εβδομάδα, πρότεινα αφού εξέτασα τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Φορέα Ελέγχου των Στοιχείων και δύο εκθέσεις Eurodac 2009 και του 2007, διάφορες τροπολογίες Δύο κατηγορίες έχουν οι τροπολογίες. Πρώτη, τεχνικές τροπολογίες. Ευθυγράμμιση συνθηνίκη της Λισαβόνας, παραπομπές στην οδηγία για τα προσόντα ή προσαρμογές διαφόρων στοιχείων του κειμένου και εσωτερικών παραπομπών. Οι άλλες τροπολογίες διευκρινίζουν το κειμένο. Μέσω παραδειγμάτων. Ας πούμε, τεχνολογία με τεχνικέ αντικαθίσει στο 4 και διευκρινίσει στο άρθρο 4-4 που αφορούν το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια μεταβατική περίοδου ή προσθήκε όσον αφορά το τμήμα με τα στατιστικά στοιχεία και διευκρινίσει όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβαση στα δεδομένα. Θέλω να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων επί προτάσεω, καθώ και απόψει για το σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ του και εισηγητή για τι πρώτε συζητήσει που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο. Πριν κλείσω, θα ήθελα να προβώ σε κάποια σχόλια όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη και οι αρχές των κρατών μελών και η Europol να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac για την πρόληψη, εντοπισμό, ε, διερεύνηση τρομοκρατικών αδικημάτων και άλλα αδικήματα. Έκανε πρόταση στο Σεπτέμβριο 2009 σχετική Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορα στοιχεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τωρινή πρόταση για τη χρήση από αυτού του φορεί των στοιχείων. Υπάρχει το ενδεχόμενο, υπάρχει δυνατότητα μόνο αν η σύγκριση των εθνικών βάσεων δεδομένων με δαχτυλικά αποτυπώματα και των, και των αυτομάτων βάσεων δεδομένων με δαχτυλικά αποτυπώματα των κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 615-2008 του Συμβουλίου, απόφαση ΠΡΟΜ, δώσει αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι περαιτέρω η πρόσβαση στα στοιχεία θα είναι δυνατή μόνο για πρόληψη εντοπισμό έρευνα τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αν υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι αυτή η σύγκριση με τα στοιχεία Eurodac θα συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη εντοπισμού και διερεύνηση εξυχνίαση τέτοιων ε, εγκλημάτων. Και μία απάντηση όσον αφορά τα θερμικά στοιχεία θα ε, θα έπρεπε να έχει μια αντιστοίχηση με τα στοιχεία Eurodac και έτοιμα οι συμπληρωματικές και αν υπάρχει αντιστοίχηση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα α, μέτρα που προβλέπονται όπως η απόφαση του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών και ε, διαφόρων πληροφοριών των ε, αρμοδίων φορέων των κρατών μελών στα πλαίσια της αμοιβαίας νομικής αρρωγής. Ήθελα να ξεκαθαρίσω τα θέματα που αφορούν το πώς οι φορείς επιβολής του νόμου έχουν πρόσβαση στοιχεία. Γιατί αυτό δεν προβλέπεται συγκεκριμένα από την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Ξέρω όμως ότι τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισαν ότι θα ήθελα να προβλέπεται αυτή η πρόσβαση στην απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέκλεισε αυτή τη δυνατότητα από την τροποποιημένη πρόταση για να προωθηθεί το πακέτο για το άσυλο και να δημιουργηθεί και η υπηρεσία, η αρμόδια που θα ασχολείται με τα θέματα. Πρέπει να διερευνηθεί όμως αυτή η δυνατότητα, κατά την άποψή μου. Αν θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες οι συνάδελφοι, μπορώ να αναφερθώ και στον κανονισμό, σε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τις δυνάμεις της τάξης. Τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 9 Δεκεμβρίου. Δεύτερη συνάντηση με τους Κιώδης είναι κάτι που επιθυμώ για να συζητήσουμε τροπολογίες και δεχόμενη ψηφοφορία προσανατολισμού μπορεί να γίνει στην ε, συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ 25-26 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ήθελαν να παρέμβουν. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Ευχαριστούμε και την κυρία Μακοβέη. Θεωρώ πως ε, το σχέδιο αυτό έκθεσης ευρεώνει την πεποίθηση στο Συμβούλιο πως ε, η Κομισιόν ε, έλαβε υπόψη τα όσα συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη νέα της πρόταση. Οπότε και από πλευράς Συμβουλίου έχουμε την εντύπωση πως σε τεχνικό επίπεδο Λίγα πράγματα πρέπει να συζητηθούν ακόμα. Μιλάμε μόνο για τεχνικές προσαρμογές. Έχουμε μια καλή βάση. Βεβαίω υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ανέφερε η κυρία Μακοβέη είναι το θέμα της πρόσβασης ε, των ε, σωμάτων ασφαλείας. Στο τελευταίο Συμβούλιο Δικαιοσύνης ε, και εσωτερικό νομίζω όλα τα κρατημέλη είπαν πως ε, ήταν απογοητευμένα ε, για το ότι δεν έκανε μια σχετική πρόταση Κομισιόν για την πρόσβαση. Πράγματι στην πρόταση του 2009 ξέρετε πως το δικαίωμα της πρωτοβουλίας ε, το έχει εντελώς η Κομισιόν και είχε πει πως είναι διατεθειμένη να το εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you. The Commission. Ευχαριστώ, η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η τρίτη πρόταση από την ε, Κομισιόν ε, που εθετήθηκε σε 11 Οκτωβρίου προκειμένου να βοηθήσουμε την Βελική Προεδρία να προχωρήσουμε ε, το πακέτο ασύλου και να καταλήξουμε σε γρήγορη συμφωνία προκειμένου να ξεκινήσει το, να το έργο της υπηρεσίας του από το 2012 και μετά έχουμε διατηρήσει τους ε, στόχους της πρώτης πρότασης να βελτιωθεί η χρήση των δεδομένων για την εφαρμογή του συνθήκης του Δουβλίνου, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων, καλύτερη λειτουργία της Eurodex στο μέλλον κλπ. Η, διαχεί... η λειτουργική διαχείριση πλέον του Eurodac απαφιέται ε, στην Κομισιόν. Επίσης περιλαμβάνεται το αποτέλεσμα των συζητήσεων του Συμβουλίου και λαμβάνεται υπόψη ε, το πρώτο νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τα καινούργια στοιχεία αυτής της ε, πρότασης, να πω ότι υπάρχουν ε, διατάξεις για την λειτουργία της επιτροπολογίας του Δουβλίνου που θα περιλαμβάνει πλέον και το, και το Eurodac θα ενημερώνονται οι αιτούντες άσυλο για τα δικαιώματά που προκύπτουν από το Δουβλίνο και το Eurodac. Ε, επίσης, ε, διευκρινίζουμε ε, θέματα τα οποία ήταν ε, εμφανίζονταν στο προήμιο και τώρα περνάνε στο διατακτικό. Μετά, η, το θέμα της πρόσβασης από τις αρχές επιβολής του νόμου ε, διαγράφεται, οπότε διαγράφονται και αντίστοιχες ε, μεταβατικές διατάξεις. Επίση υπάρχει κι άλλο ένα θέμα που είναι σχετικό με μελλοντικέ διαπραγματεύσει ενδεχομένων. Πρέπει να συμφωνήσουμε επί αυτού. Είναι το θέμα τη περίοδου αποθήκευση ε, δεδομένων κατηγορία 2. Δηλαδή παράνομη παράτυπη εισόδου. Ε, άτομα τα οποία συλλαμβάνονται κατά την παράνομη διέλευση εξωτερικών συνόρων. Όπω θα θυμάστε, στον ισχύοντα κανονισμό αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται για δύο χρόνια, αλλά η Κομισιόν ήδη από την πρώτη πρότασή τη ε, ε, και τώρα βέβαια, προτείνει χαμηλότερη περίοδο, ενό έτου συγκεκριμένα, προκειμένου να είμαστε συνεπείς με τον, το στόχο του κανονισμού του Δουβλίνου. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η DPS ε, έχουν διαφορετική άποψη από το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Τώρα, το θέμα της ε, πρόσβασης, η Κομισιόν ε, σημειώνει την προτίμηση ορισμένων κρατών μελών να ξαναμπεί το θέμα στην πρόταση. Η Επίτροπος έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών, είπε ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί αλλά μόνο ως τμήμα μιας ευρύτερης, πιο ισορροπημένης πρότασης και μιας πιο επικοδομητικής στάσης του Συμβουλίου για το όλο πακέτο ασύλου. Ευχαριστώ. the... ε, ξεκινάμε τη συζήτηση. Έχω αρκετούς ομιλητές. Ξεκινάμε τον κύριο Μωράης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το κεντρικό σημείο ήταν το θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα πλευράς ε, ε μονα, ε, υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Τώρα η απόσυρση αυτού του σημείου μας δίνει την δυνατότητα να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και βέβαια να υποστηρίξουμε και ε, πολλές από τις τεχνικές ε, τροπολογίες που προτείνει η κυρία Μακοβέη. Πρόκειται για μια αναδιατύπωση, ε, συνεπώς περιοριζόμαστε σε τροπολογή, τροποποίηση των πτυχών που έχει τροποποιήσει η Κομισιόν στην αναδιατύπωση. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με την κυρία Μακοβέη και νομίζουμε ότι ακολουθεί μια πολύ σόφρονα στάση το βασικό εμπόδιο το αφαίρεσε η Κομισιόν που ήταν η πρόσβαση. Ε, συνεπώς ε, νομίζω ότι πάμε καλά. Η Βελική Προεδρία προχωράει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σκιώδης μας η κυρία Λάτφορντ δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα, οπότε θα μιλήσω εκ μέρους της. Αλλά αυτά που ήθελε να πει αντικατοπτρίζουν στις απόψεις της Άλντε. Θα ήθελα να υποστηρίξουμε την έκθεση Μακοβέη και κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν για καλύτερα πρότυπα χαιρόμαστε που ελήφθησαν υπόψη και συμπεριλήφθησαν στην έκθεση. Υποστηρίζουμε επίσης το ότι η έκθεση αυτή τη στιγμή αντικατοπτρίζει το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει άρρητη δυνατότητα τα κράτη-μέλη οι δυνάμεις της τάξης των κρατών μελών έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, ακούγοντας αυτά που μας είπε η συγγήτρια και τα όσα είπε και το Συμβούλιο, πρέπει να τονίσουμε ότι προβληματιζόμαστε όσον αφορά το περιθώριο που έχει αφαιθεί για μελλοντική αλλαγή αυτού του γεγονότος Ακούσαμε το Συμβούλιο να μας λέει ότι θέλει να επιτρέψει την πρόσβαση από πλευράς δυνάμων της τάξης στην βάση δεδομένων και είμαστε κάθετα αντίθετοι. Και είναι ένα ισχυρό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς το Συμβούλιο, προς τη Βελική Προεδρία, προς την Ουγγρική Προεδρία και για πολλούς λόγους έχουμε αυτή τη στάση. Νομίζω ότι όλοι τις τελευταίες εβδομάδες λάβατε κάποιες προειδοποίησεις από αρχές προστασίας των δεδομένων και από φορείς κοινωνίας των πολιτών που ετέθησαν κατά της προτάσεως λόγω αυτής της πρόσβασης που θα παραβίαζε ε, τους περιορισμούς και θα μετέτρεπε το Eurodax σε ένα εργαλείο εξυχνιάσεως εγκλημάτων και αυτό ε, θα παρέμβει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εφόσον οι δυνάμεις της τάξης θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν και άλλα βιογραφικά ε, ε, στοιχεία που συνδέονται με τα θηλυκά αποτυπώματα. Και αυτό είναι κάτι που απορρέει από την ανάλυση συνεπιών του 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό σημαίνει ότι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουμε αύξηση του κόστους λόγω της αυξημένης κατεργασίας στοιχείων του Eurodac. Ελπίζουμε το Συμβούλιο λοιπόν να μην θέλει να ξεκινήσει την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου που θα είναι πολύ δαπανηρό και δίνει υποστηθέμενη αξία αμφισβητήσιμη και δεν συνάδει με τους σκοπούς λειτουργίας της υπηρεσίας. Ελπίζουμε να κλείσει αυτή η ανοιχτή πόρτα που παραμένει αυτό το περιθώριο. Ευχαριστώ Ρενάτε. Ο κύριος Ντεγιόγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καμιά φορά εκπλήσωμαι Βλέπω ότι λείπει το ιστορική μνήμη από κάποια κράτη-μέλη. Αν δουν τα αρχεία τους και δουν τι έλεγε η σύμβαση του Δουβλίνου, ήταν η σύγκριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για να το υπεύθυνο για το αίτημα υποβολής ε, ασύλου. Ποτέ. Ποτέ προευλήθη το επιχείρημα να χρησιμοποιηθούν τα αποτυπώματα κατά το εγκλήματος της τρομοκρατίας. Θα, ε, θα παραβιαστεί η προστασία των δεδομένων να ακολουθηθεί αυτή η μεθοδό, αν αλλάξει ο σκοπός χρήσεως ενός μέσου, δίνοντας πρόσβαση στις δυνάμεις της τάξης ε, στα δαχτυλικά αποτυπώματα της Eurodac. Είναι σοβαρή παράβαση αυτή. Και ανακουφίστηκα που έβγαλε αυτή την πρόβλεψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δυνάμεις τάξης δεν έχουν πρόσβαση. Στο Συμβούλιο βλέπω ότι συζητείται όμω η επανεισαγωγή αυτής της δυνατότητας. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ ασφαλμένο και λάθο μήνυμα. Και νομικά θα δημιουργούνται πολλά προβλήματα με αυτό το εργαλείο. Απ' την άλλη συμφωνώ με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το πακέτο του ασύλου. Τέλος. Ευχαριστώ τη Μόνικα Μακοβέη για τις τεχνικές τροπολογίες που αφορούν την έκθεση και για τις τροπολογίες που πρότεινε. Νομίζω ότι η συζητήσεις θα είναι καρποφόρες. Όμως ε, παρατηρώ ότι στην έκθεση της Μακοβέ υπάρχει αναφορά στην πρόσβαση από πλευράς των δυνάμεων της τάξης. Λυπούμε που υπάρχει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άρμπρεχτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιοδησηγητές για την προσέγγιση που είχαμε μέχρι τώρα και να πω πως υποστηρίζω την κυρία Βέμπερ για το θέμα της ε, πρόσβασης ε, των δυνάμεων της τάξης. Είχαμε έντονη κριτική από πλευράς Κοινοβουλίου και αναφέρθηκαν πολλά επιχειρήματα ε, για το γιατί δεν είναι αναλογικό να ανοίξουν οι νέες αυτές βάσει δεδομένων για τις δυνάμεις της τάξεως. Οπότε θα ήθελα η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν για την πρόταση αυτή. Αλλά από ό,τι ακούω αυτό το στηρίζει ομόφωνα το Συμβούλιο, οπότε θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Και νομίζω πως θα είναι κρίσιμο να ξεκαθαρίσετε στο Κοινοβούλιο εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Thank you. Monica. Uh, thank you. So it's, it's... Monica. Ε, ευχαριστώ. Είναι σαφές αυτό το οποίο, μετά από αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν και το Συμβούλιο, πώς θα συνεχίσουμε με την πρόταση ως έχει. Και το Συμβούλιο θα κάνει μια πρόταση για πρόσβαση των υπηρεσιών ασφαλείας. Οπότε έχω καταλάβει όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες είναι σαφείς και εν ειρήνη. Ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας. Δεκτή η προθεσμία και θα συζητήσουμε στην επόμενη συζήτηση τα της πρόσβασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μόνικα. Μια που είναι ήδη εδώ η κυρία Μάλμστρομ, η Επίτροπος, προτείνω να ξεκινήσουμε το σημείο 16 τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας να ακούσουμε την κυρία Επίτροπο και το 14 και 15 για την ε, Βραζιλία να τα δούμε μετά. Το θέμα είναι εάν οι συγγήτρες η κυρία Μακοβέη και ο κύριος Έντσιου συμφωνούν. Να ακούσουμε πρώτα την Επίτροπο και μετά να συνεχίσουμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Οπότε θα δώσω λόγο στην κυρία Μόναστρα μου. I'm very happy to receive... Χαίρομαι που καλωσορίζω την Επίτροπη κυρία Μάλστρομ που θα μας ε, παρουσιάσει την ε, <clears throat> ανακοίνωση Επιτροπής για την ε, <clears throat> ε στρατηγική εσωτερική ασφάλιση Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη, πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. <clears throat> Δημοσιεύθηκε την προηγούμενη Δευτέρα. Η Επιτροπή μας θα υιοθετήσει μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία με συγκεκριμένα την κυρία Μπορσαλίνο για το θέμα τη εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την διαθεσιμότητά σα και την προθυμία σα, κύριε Μάλστρομ. Σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μια ακόμα φορά. Συναντώ Έχω συναντήσει πολλούς ε, και πολλές από εσά ε, τις τελευταίες εβδομάδες ε, επανειλημμένως για διάφορα θέματα. Σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ τη Γραμματεία και την Προεδρία που αλλάξατε λίγο την σειρά των θεμάτων στη μερίσια διάταξη. Έτσι καθίστατε δυνατό να σας παρουσιάσω αυτή την ανακοίνωση πριν την παρουσιάσω στο Συμβούλιο. Πάντοτε καλό αυτό. Υιοθετήθηκε από την Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα αυτή η ανακοίνωση και εκφράζει την βούλησή μας να δούμε την ασφάλεια σε με πιο ολιστικό τρόπο και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τα οποία μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πολλοί από εμάς ε, δεν ήταν ικανοποιημένοι που στο παρελθόν που η ασφάλεια ε, είχε κατακαιρματιστεί. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια ε, να ακολουθήσουμε μια άλλη προσέγγιση, ε, μια πιο ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα, τις προκλήσεις με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Έχουμε εντοπίσει πέντε θέματα, πέντε τομείς ε, που χρειάζεται να δράσουμε. Βέβαια η ασφάλεια είναι η αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προσθέσουμε αξία. Οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, διαχείριση εσωτερικών συνόρων και ε, ε, ανθρωπογενείς καταστροφές. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε την ασφάλεια των ατόμων και των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στην Ευρώπη. Ξεκινώντας από το πρώτο ζήτημα, ας ξεκινήσω από το οργανωμένο έγκλημα, γνωρίζουμε ότι ε, πολλά πτέσματα τα οποία βλέπουμε ε, στην καθημερινή ζωή, κλοπές αυτοκινήτων ε, κλπ. αποτελούν τμήμα ενός δικτύου οργανωμένου εγκλήματος. Οπότε πρέπει να επιτρέψουμε στις ε, αρχές της τάξης να μπορούν διασυνοριακά να ε, διώκουν, να καταδιώκουν ε, τέτοιου είδους δίκτυα, κυρίως μέσω της Παρακολούθηση του, της ροής του, του χρήματος. Είναι το πιο ευαίσθητο του ε, σημείο. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα από παράνομες δραστηριότητες δεν ε, θα ε, νομιμοποιούνται στην κανονική νόμιμη οικονομία. Πώς μπορούμε να κατάσχουμε περιουσιακά στοιχεία και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε καλύτερα τη διαφθορά και την νομιμοποίηση παρανόμων προσόδων. Αυτές είναι οι προτάσεις οι οποίες θα υποβάλουμε την άνοιξη. Για την τρομοκρατία. Γνωρίζουμε δυστυχώ ότι η Europol ε, ανέφερε περίπου 300 ε, τρομοκρατικές πράξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι. Ε, τις τελευταίες ε, είδαμε κάποιες από αυτές τις πράξεις στα φορτία που ερχόντουσαν από την Ιεμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Επίσης έχουμε κάποια κομμάτια της ε, κοινωνίας μας τα οποία αποκόπτονται από την υπόλοιπη κοινωνία και είναι εύκολα θύματα των ε, ε, στρατρολόγησης από πλευράς τρομοκρατών. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε προτάσεις για την πολιτική ασφάλειας και θα προσφέρουμε μια ε, πλατφόρμα για την αποφυγή του της, ε, ε, της αύξησης του ευάλωτου ε, κομματιών ε, τμήματων του πληθυσμού μας. Επίσης του χρόνου θα προβάλλουμε πρόταση ε, για τα στοιχεία TFTP και το πώς μπορούμε να σας τα παρουσιάσουμε. Ε, σε ό,τι αφορά το, το στον κυβερνοχώρο, ε, ε, δεν χρειάζεται κανείς να επιτεθεί εναντίον πυρηνικών σταθμών για να τελέσει τέτοιου είδους αδικήματα. Ε, μπορεί να γίνει και μέσω αφαίρεσης ποσών ηλεκτρονικά από λογαριασμούς κλπ. Νομίζω ότι όμως η οι ε, τρομοκράτες μπορούν να κάνουν και τα δύο και να επιτεθούν εναντίον υποδομών και να κλέψουν χρήματα. Οπότε ε, χρειάζεται ένα δίκτυο ε, ομάδων άμεσης ε, δράσης για εγκλήματα κυβερνοχώρου σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν είναι καλά προετοιμασμένα για αυτό το θέμα, για την αντιμετώπιση τέτοιου είδου εγκλημάτων. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να είμαστε πιο έτοιμοι σε έναντι μελλοντικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Όπως γνωρίζετε έχουμε προτείνει επίσης να γίνουν, καθαστούν εγκλήματα, αδικήματα, τα botchnets. Ε, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων χρειάζεται περισσότερο συντονισμό, έτσι ώστε εκεί που είναι τα θερμά σημεία των εξωτερικών συνόρων, οι συνοριοφύλακε να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ του και να αντιμετωπίζουν ε, όλων των ειδών τη ε, παράνομε Του χρόνου θα υποβάλουμε προτάσεις για το σύστημα επιτήρησης εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το λαθρεμπόριο παρανομών αγαθών, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη βάση για συνεργασία στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις και τις ε, θεομηνίες, ε, την περασμένη περασμένο μήνα ε, είδαμε κάποιες ε, τρομακτικές τέτοιου καταστροφές, ε, έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία, παράδειγμα, δημιούργησε πολλά προβλήματα ε, οι πλημμύρες στην ε, Μαδέρα, ε, τοξικά απόβλητα στην Ουγγαρία. Όλες αυτές οι καταστροφές απαιτείται να αντιμετωπιστούν από κοινού. Είναι διάφοροι τομείς που θα πρέπει να συνεργαστούν. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλισης μεταφορών, όχι μόνο οικονομικό θέμα, όχι μόνο χρηματοπιστωτικό θέμα. Είναι, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μαζί. Χρειάζεται ένα σύστημα ε, αντιμετώπιση κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να αναπτύξουμε μελέτες αξιολόγησης ε, κινδύνου ε, έτσι ώστε ε, να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπιση κρίσεων. Συνεργαζόμαστε και με πολλούς άλλους επιτρόπους. Είναι μια διαδικασία στην οποία χρησιμοποιήσαμε τι απόψει τη δικέ σα, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κρατών μελών, ανθρώπων που εργάζονται με τέτοιου είδου ζητήματα και από όσο ε, γνωρίζω η κυρία Μπορσελίνο θα είναι εισηγήτρια για μια ε, εισήγηση πρωτοβουλία την οποία ετοιμάζεται. Πολύ ευχαριστώ θα δούμε μετά ε, τις συστάσεις σας. Γιατί δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, δεν, ε, δεν πρέπει να παραμείνει ένα ακόμα ε, χαρτί αυτή η ανακοίνωση, έχουμε προκλήσεις μπροστά μας και θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι ε, τις γνωρίζουμε και ότι εργαζόμαστε προκειμένου να, να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις ζημιές. Θα αξιολογήσουμε την πρόοδο μέσω μιας ετήσιας ε, έκθεσης με συστάσεις για περαιτέρω δράσεις και αυτή η δημοσίευση αυτή τη ετήσια έκθεση ε, θα είναι ευκαιρία να συζητάμε και με εσά και με το Συμβούλιο για τέτοιου ζητήματα. Αυτή είναι η στρατηγική μα για την ε, βελτίωση τη εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, την αναπτύξαμε μαζί με εσά και με το Συμβούλιο. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε στο μέλλον στενά για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Αυτά είναι μια πολύ συνοπτική παρουσίαση αυτού του μακροσκελούς και σημαντικού εγγράφου. Είμαι στη διάθεσή σας και σήμερα και οποιαδήποτε άλλη στιγμή όταν αρχίσουμε να ε, εργαζόμαστε για καθένα από αυτά τα ζητήματα χωριστά. Ευχαριστώ. Το εκτιμούμε το ότι ήρθατε και ότι ήρθατε σε εμά πρώτοι. Πρώτα μάλλον. Έχω το κατάλογο αγορητών. Να δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Μπορσαλίνο, την εισηγήτρια. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω αν ακούτε τη φωνή μου. Έχω σχεδόν χάσει τη φωνή μου. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα την Επιτρόπο, την κυρία Μάλστρομ, που ήρθε να μας παρουσιάσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη και την εσωτερική ασφάλεια. Πολύ σύντομα στην πρώτη ανταλλαγή απόψε, να επαναλάβω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συμβάλλει και να παίξει το ρόλο του στην επεξεργασία μια στρατηγική που έχει σκόπο να αποφύγει και να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Πέρα από τους στόχους που αναφέρονται στην ανακοίνωση, θα ήθελα μεθοδολογικά να ληφθούν υπόψη κάποιες πτυχέ για να ξεπεράσουμε πέρα από αυτά που αναφέρονται στην ίδια την ανακοίνωση. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ποιο πραγματικό κίνδυνο ελοχεύει για την Ευρώπη δεν αρκεί να πούμε ότι τέσσερις από τους πέντε Ευρωπαίους ανησυχούν. Χρειάζεται πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για να δούμε την πραγματική εμβέλεια της απειλής. Μιλώ για τα στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα, για την ανακύκλωση ελεύθερης του χρήματο, για το προϊόντα της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια μέσα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και εδώ θα πρέπει να γίνει μια ακριβή απογραφή και με ποιο τρόπο η Europol και το Eurojust και το Frontex μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους μετά πιστεύω είναι σημαντικό να εμπλακούν και άλλοι φορείς στη διαμόρφωση στρατηγικής, όπως τα Εθνικά Κοινοβούλια και άλλοι εθνικοί φορείς, όπως οι δικαστές, η κοινωνία των πολιτών, οι ενώσει που σε τοπικό επίπεδο ασχολούνται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στις καλές εθνικές πρακτικές, αυτές που λειτουργήσαν επιτυχώς και μετά θα πρέπει να εξαχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη στιγμή που θα έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία, και περάσει αυτά τα στάδια πρέπει να καταλάβουμε τι λείπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώ πραγματικά μπορούμε να αντισταθούμε στο οργανωμένο έγκλημα και στην τρομοκρατία. Βεβαίω είμαι έτοιμη να ακούσω και να δεχτώ προτάσει των συναδέλφων και εύχομαι καλή εργασία σε όλου. Σα ευχαριστώ κύριε Μπορσαλίνο. Κύριε Λαμπρινίδη, έχετε το λόγο. Thank you very much. for Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Επίτροπε. Δύο παρατηρήσεις έχω Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά πιέζει ο χρόνος. Γι' αυτό το πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Το ένα αφορά το τι γίνεται στο διαδίκτυο και το τι, προσπαθούμε, το τι εγκλήματα προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και το άλλο φορά βεβαίως την ε, ριζοσπαστικοποίηση. Βεβαίως όλα αυτά σχετίζονται με τον ορισμό. Τι είναι η ιστορική ασφάλεια, πώς ορίζεται, έχουν αίσθηση πως προσπαθείτε εδώ πέρα να πιάσετε όλα αυτά με ένα τεράστιο δίχτυ. Δηλαδή όποιος βγάζει χρήματα από οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό, καλύπτεται. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Ανησυχώ ιδιαίτερα πως αναφέρεται ερητός και στην ανακοίνωση αυτή που μιλάτε για την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ως θέμα εσωτερικής ασφαλείας. Καταλαβαίνω πως δεν το είπατε στην ε, παρουσίασή σας πώς ε, μιλάτε για το ηλεκτρονικό έγκλημα όταν επιτίθεται σε κρίσιμες υποδομές, ε, όταν χρησιμοποιείται για εμπορία παιδιών, αλλά γιατί δεν αναφέρεται η εμπορία παιδιών και υπάρχει με παχιά γράμματα η παραβίαση της ε, πνευματικής περιουσίας. Είναι σημαντικό ζήτημα, θα το συζητήσει το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια σύσταση. Αλλά φτάνει στα όρια της φαντασίας ε, το πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει προτεραιότητα της στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας. Εκτός να ορίσουμε την εσωτερική ασφάλεια τόσο ε, ευρύτατα ώστε να πούμε πως οποιοδήποτε δίκτυο βγάζει χρήματα, έστω και αν δεν πηγαίνουν στον, στην τρομοκρατία, το αντιμετωπίζουμε. Ανησυχώ, δεν θέλω να μπει εδώ πέρα, ούτε θέλω σε οποιαδήποτε πολιτική της Κομισιόν να μπαίνει αυτό εδώ μέσα. Δεύτερον, για τη ριζοσπαστικοποίηση. 26 Απριλίου έβγαλε μια επικίνδυνη, θεωρώ εγώ, ανακοίνωση το Συμβούλιο. Αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό για να συλλέξουν πληροφορίες από τα κράτη-μέλη με βάση ένα ερωτηματολόγιο για την ριζοσπαστική ιδεολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζουν, δεν εξηγούν τι, ποια είναι αυτή η ακραία ιδεολογία Δηλαδή σχεδόν επιτρέπουν να μπει στην κατηγορία αυτή οτιδήποτε. Υπήρχε μια ακραία πολιτική άποψη που δεν μας αρέσει. Ζητάνε πληροφορίες οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν και τους γείτονε, τους φίλους και τους συγγενείς των υπόπτων, των ανθρώπων που υποπτεύονται οι αρχές. Και δημιουργούν γενικώ μία βάση δεδομένων, η οποία είναι τεράστια, δεν ορίζεται, δεν ορίζεται η νομική της βάση και κατά την άποψή μου είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη. Η Κομισιόν κάνει τίποτα για να συντονίσει ή να εφαρμόσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτό το μηχανισμό συλλογής δεδομένων για τη βάση δεδομένων. Εάν όχι το έχετε παγώσει ή το έχετε σταματήσει, ξέρετε τι κάνει το Συμβούλιο εδώ πέρα. Γιατί και πάλι το πώς ορίζουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και την ιδεολογία, ε, το θέμα του ορισμού δηλαδή μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες για την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σταύρο. Η κυρία Ίνετφέλτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, καλώς ορίζω την ολοκληρωμένη αυτή, όπως είπατε, προσέγγιση. Νομίζω πως ώρα ήτανε. Συμφωνώ και θεωρώ πως το κοινοβούλιο μας ε, οπωσδήποτε θα συνεισφέρει στη συζήτηση, αλλά όπως και ο Σταύρος θεωρώ και εγώ πως χρειάζεται περισσότερη συζήτηση για τους ορισμούς, για τις αρχές, για τους στόχους, γιατί πρώτα απ' όλα θεωρώ πως ε, ένα από τα πράγματα τα οποία λείπουν εδώ πέρα και οπωσδήποτε στον τομέα που με απασχολεί εμένα, την καταπολέμηση της δημοκρατίας, είναι τα στοιχεία, τα γεγονότα, η αξιολόγηση του χρόνου θα έχουν περάσει 10 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Ε, ευρύτατα μέτρα έχουν ληφθεί, έκτοτε σωστά λέτε πως δεν είναι και πολύ συνεκτικά μέτρα, αλλά μικρή ιδέα έχουμε για το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων. Έχουμε κάποια ιδέα για το τι επίπτωση έχουν ε, στις ε, πολιτικές ελευθερίες, αλλά λίγα πράγματα για το κόστος ξέρουμε. Οπότε για οποιαδήποτε μέτρο ε, θα πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα μια εικόνα του πού είμαστε αυτή τη στιγμή και το τι χρειάζεται. Δηλαδή να δούμε πού χρειάζονται οι δυνάμεις επιβολής τάξεως νέους σπόρους και μετά. Γιατί καμιά φορά πολεμάμε ανεμόμυλους και επηρεαζόμαστε τόσο πολύ στην εποχή μας από τις εικόνες και τη φαντασία. Πρέπει λοιπόν η πολιτική μας να βασίζεται στα γεγονότα. Κάποια άλλα συγκεκριμένα ζητήματα. Χαίρομαι που συμπεριλάβατε την κλοπή της ταυτότητας στο κεφάλαιο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, γιατί μιλάμε εδώ πέρα για ένα ε, από ε, του ταχύτερα αναψώμενους τομεί του εγκλήματο και βεβαίω αφορά άμεσα του πολίτε μα. Και όμω, ε, ενώ είναι χρόνια στο προσκήνιο, τα κράτη-μέλη αρνούνται να το αντιμετωπίσουν, γιατί δεν θέλουν να προσαρμόσουν του νομικού ορισμού κλοπή ταυτότητα έτσι ώστε να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό ορισμό. και όλοι ξέρουμε πω εάν υπάρχει ένα έγκλημα το οποίο είναι πραγματικά διεθνές είναι αυτό Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τέλος δημιουργήσαμε τεράστιες νέες εξουσίες για, δημόσιο, για τις δημόσιες αρχές για να ελέγχουν τους πολίτες. Αλλά οποιοδήποτε νέο μέτρο, οποιαδήποτε νέα εξουσία που δίνουμε στις αρχές θα πρέπει να αντισταθμίζεται από νομικές δικλείδες ασφαλείας για τους πολίτες. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κοινό και πρέπει να πηγαίνει μία και μία. Δηλαδή νέα εξουσία, νέα διασφάλιση. Γιατί μιλάμε για τα προσωπικά δεδομένα. Ο τεράστιος αριθμός βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί για λόγους ε, τάξης και ασφάλειας είναι μάνα εξ ουρανού για όσους θέλουν να κλέψουν την ταυτότητα κάποιου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν θέλουμε να δώσουμε απαραίτητες νέες εξουσίες, κάθε νέο μέτρο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μια δικλίδα προστασίας των πολιτών. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Ζεκολίνο. Μεγάλη χαρά που συναντούμαστε μαζί σας κυρία Μάλστρομ για μια ακόμη φορά. Χρήσιμη συζήτηση για το Κοινοβούλιο όπως σίγουρο πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμη και για σας. Αυτή η ανακοίνωση, όπως όλες οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροφής, δείχνει κάποια στοιχεία προβληματισμού σοβαρού και δίνει τη δυνατότητα και στο Κοινοβούλιο μας Επιτροπής Ελευθεριών να προτείνει κάποιες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Θα ήθελα να σταθώ κυρίως στο τμήμα εκείνο της παρέμβασης που αφορά το οργανωμένο έγκλημα και την αντίθεσή του στο οργανωμένο έγκλημα. Πρώτη πτυχή λοιπόν. Η κατάσχεση των αγαθών της μαφίας, των οργανωμένου εγκλήματος, της αφαιρέσεως των αγαθών του οργανωμένου εγκλήματος, ε, απλούστευση των διαδικασιών χρειάζεται για να επιτευχθεί μια ταχεία χρησιμοποίηση αυτών των αγαθών που κατάσχονται το οργανωμένο έγκλημα για να επενδυθούν αυτά τα αγαθά κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Και όπως και στην Ιταλία δεν χρησιμοποιείται πολύ καλά αυτό το που κατάσχεται από τη μαφία, διότι είναι πολύ δυσκίνητες οι διαδικασίες και δεν επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της χρήσεως των αγαθών αυτών μέσω πλούστευσης. Και μετά η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τον Ιούνιο του 2010 στο Παρίσι κατόπιν πρότασης του Γάλλου Υπουργού ξεκίνησε μια προσπάθεια κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ένα σύμφωνο με συγκεκριμένους προσανατολισμούς θα πρέπει να απτυχθούν βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σε αυτό το κοινοβούλιο δεν είναι απλό κάτι τέτοιο, δεν είναι απλό να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που αφορούν τα ναρκωτικά, την ε, εξάρτηση από τα ναρκωτικά κλπ. Και ζητώ από την Επίτροπο, την κυρία Μάλστρομ, αν επ' αυτού του θέματος τις προτάσεις του Γάλλου Υπουργού αν υπάρχει κάποια σκέψη, κάποιος προσανατολισμός και αν θα προωθήσετε κάτι σχετικά με αυτό το θέμα και στα πλαίσια της ανακοινώσεως που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστώ. Και τώρα θα στραφώ προς την κυρία Επίτροπο. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και μετά θα ακολουθήσει άλλος ένας γύρος. Έχουμε έξι ακόμα συναδέλφους που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο, Κύριε κύριε Σίπαλ, Σβίμπαρ, Άλμπρεχτ, ο κύριο Μόλτερ, η κυρία Μπλινκεβιτσιούτε και η κυρία Χάνκες. Και η κυρία Γκρίσμπεκ. Δεν θα έχουμε το χρόνο όμως. Λίσμπεκ, Ρομέρο Λόμπες και Σίρφελ σας αναφέραμε θα τα καταφέρουμε. Κυρία Ένστ, και εδώ κλείνει ο κατάλογος των αγορητών. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για το πολύ ενδιαφέρον που δείχνετε. Καλό αυτό για μελλοντικές συζητήσεις. Προς την κυρία Μπορσελίνο. Ελπίζω να βελτιωθεί η φωνή σας, ο καιρός δεν βοηθάει βέβαια. Ε, εξετάζουμε το εξής. Δεν προτείνουμε πολλά καινούργια ε, μεγαλόσχημα νομοθετικά κείμενα. Εξετάζουμε τι υπάρχει, αν λειτουργεί, αν, μπορεί να, αν πρέπει να βελτιωθεί, ε, τι έμπνευση μας δίνουν ε, οι εθνικές νομοθεσίες, για παράδειγμα το πάγωμα ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Πολλοί από εσά έχετε σε εθνικό επίπεδο ε, δουλέψει πολύ με αυτό το θέμα. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από όλα αυτά τα νομοθετικά κείμενα που υπάρχουν αυτή τη ε, στιγμή οι αστυνομικοί λένε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία που υπάρχει δεν λειτουργεί. Πρέπει να δούμε γιατί δεν, γιατί δεν λειτουργεί. Οι εγκληματίε ε, μετακινούν ποσά μέσω διαμέσου των συνόρων και πρέπει να μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Αυτό θα το κάνουμε του χρόνου και θα πρέπει να συνεργαστούμε εσά. Κύριε Λαμπρινίδη, πολλά πράγματα δεν έχουμε συμπεριλάβει γιατί υπάρχουν πολλέ παράλληλε πρωτοβουλίες που λαμβάνει χώρα. Ε, καταλαβαίνω ότι η παρενόχληση παιδιών είναι πολύ σημαντική, λοιπά. Η, ε, η πνευματική διοκτησία περιλαμβάνεται μόνο αν έχει σχέση με το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, καμία σε άλλου τύπου. Ε, επίσης δεν προσπαθούμε ε, να δημιουργήσουμε κανόνε είδου βάση δεδομένου οτιδήποτε άλλο. Εμείς απλώς ανταποκρινόμαστε στο αίτημα των τοπικών αρχών να υπάρχουν πλατφόρμες, κοινές πλατφόρμες διότι πολλοί προσπαθούν να εντοπίσουν τις δικές τους εθνικές ε, τρομοκρατικές ε, ομάδες και συνεργάζονται με άλλους, με άλλες ε, Ομάδε που εργάζονται με την ίδια κατεύθυνση, προ την ίδια κατεύθυνση κλπ. Συνεπώς δεν υπάρχει κανό είδου βάση δεδομένων, υπάρχουν πλατφόρμες μέσα στις οποίε θα μπορούν οι ε, τοπικές αρχές και ερευνητέ να ε, επικοινωνούν. Κυρία Ιντβελτ, συμφωνώ μαζί σα ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό που έχουμε και το προσπαθήσαμε ε, με τον απολογισμό για τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας που υποβάλαμε πριν το καλοκαίρι. Και σίγουρα όταν προτείνουμε κάτι καινούριο, ε, οποιοδήποτε καινούριο μέτρο, ε, θα το ισορροπούμε με ε, εγγύσεις. Βέβαια, τα κράτη-μέλη έχουν τις δικές τους πληροφορίες. Εμείς δεν έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που είναι μυστικές και θα μας χρησιμεύαν ε, αλλά σύμφωνα με τα όσα έχουμε θα οικοδομήσουμε και το, τις προτάσεις μας. Οποιαδήποτε πρόταση από δική σας πλευράς βέβαια ε, θα λαφθεί υπόψη και οποιαδήποτε δική μας πρόταση θα ακολουθείτε από μέτρα προστασίας του πολίτη. Ε, <clears throat> σε ό,τι αφορά την ε, κλοπή ταυτότητας πράγματι είναι ένα σημαντικό ε, θέμα. Εγώ έχω πολλού ε, φίλου που έχουν υποστεί τέτοιου είδου ε, ενέργειες και επίση κλοπή χρημάτων από λογαριασμού κλπ. θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Τζακολίνο, η πρόταση αυτή του Γάλλου Υπουργού υποβλήθηκε πέρσι την άνοιξη, την προηγούμενη άνοιξη μάλλον. Και την επόμενη άνοιξη θα υποβάλουμε μια έκθεση πρόοδου, να δούμε πού βρισκόμαστε. Σίγουρα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι πολύ σημαντικό. Εξε... Ετοιμάζουμε, ε, επεξεργαζόμαστε μεθόδους ε, οι οποίες θα το αντιμετωπίσουν. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος γύρος, η κυρία Σίπερ, Σβίπερ, Άλμπρεχτ, ο κύριος Μόλτερ και η κυρία Μπινκεβιτσιούτε. Και μετά ο τελευταίος γύρος, η κυρία Ζίμπερ είναι πρώτη. Dank. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη σύνοψη αυτού του εγγράφου και τη σύνταξή του γιατί θέλαμε να δούμε όλες αυτές τις πτυχές των νομοθετικών προθέσεων. Τώρα για την πτυχή εσωτερικής ασφάλειας και καταπολέμηση του τρομοκρατίου, της τρομοκρατίας συζητάμε και με ανταλλαγή δεδομένων αλλά και για τα τεχνικά ζητήματα όπως τους ε, σκάνερ, ε, τους ολόσωμους και χαίρομαι για το ότι πλέον μιλάμε για την πρόληψη, για το τι σημαίνει ριζοσπαστικοποίηση, πού στρατολογούνται οι πιθανοί δράστες και το τι μπορεί να γίνει ε, από κοινού με τα κράτη-μέλη και νομίζω είναι σημαντικό αυτό, όπως επίσης και η αναγνώριση του γεγονότος πως οι δράστες δεν προέρχονται μόνο από τρίτες χώρες, αλλά και ε, στρατολογούνται εντός της Ένωσης, δεν πρέπει να το παραμελούμε αυτό. Στο θέμα ενός ευρωπαϊκού συστήματος PNR δεδομένων αεροπορικών επιβατών ε, είμαι επιφυλακτική γιατί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως των μελιωδών ε, ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό το θέμα αυτό ούτως ή άλλως αποτελεί αντικείμενο στενής συνεργασίας και μιλάμε για ανταλλαγή δεδομένων και δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ποια επιπρόσθετη αξία θα έχει ε, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω πως θα ξεκαθαρίσει αυτό ούτως ή άλλως στη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επίτροπο την κυρία Μάστρον που ήρθε σήμερα για να μας μιλήσει για τη στρατηγική αυτή. Είναι πάρα πολύ καλή αφετηρία. Πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και πρέπει να εκφράσουμε και τις ανησυχίες μας για πολλά ζητήματα. Τα περισσότερα που ήθελα να πω καλύφθηκαν ήδη από το Σταύρο και από τη Σοφή. Και εγώ έχω πρόβλημα στον αφορά τον ορισμό της εσωτερικής ασφάλειας και για μένα η ασφάλεια του Ευρωπαίου πολίτου είναι το σημαντικότερο. Όμως έχουμε διαφορετική αντίληψη. Τώρα μιλάμε για εσωτερική ασφάλεια, έχουμε εθνική ασφάλεια, μιλάμε για ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, πολλά από αυτά θα καλυφθούν από τη στιγμή που θα μας κατατεθεί κάθε πρόταση. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω ότι κατανοώ ότι τέσσερις στους πέντε πολίτες ανησυχούν όσον αφορά την ασφάλειά τους. Θέλουν καλύτερη ασφάλεια. Το ότι όμως θεωρούν ότι μπορούν να απεμπολίσουν τα δικαιώματά τους δεν με εντυπωσιάζει πολύ διότι αφορά το πόσο ενήμεροι είναι οι πολίτες και νομίζω ότι η δική μας δουλειά είναι να προστατεύσουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις αξίες μας, τις παραδοσιακές πολιτικές ελευθερίες. Συμφωνώ απόλυτα, όσο πιο σκληροί θέλουμε να είμαστε για την προστασία της ασφάλειας, τόσο πιο σκληροί πρέπει να γίνουμε ταυτόχρονα για την προστασία των νομικών έχει εγγύων και των δικαστικών αποζημιώσεων ε, για τους πολίτες. Ευχαριστώ κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσετε τον κανόνα ότι στο πρώτο γύρο όλες οι ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο και να εκφράσουν την άποψη της ομάδας, γιατί οι πράσινοι και οι γκουε δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Θα ήθελα αυτό να το τηρούμε. Επίτροπε Μάλστρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας υποβάλατε με τέτοια πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ποιοι είναι οι στόχοι μας και να συζητήσουμε λεπτομερείς προτάσεις. Και όχι απλώς θεωρίες αφηρημένες, ασφάλεια, θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Είναι σημαντικό να μπαίνουμε στις λεπτομέρειες. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν σαφείς ορισμοί, όπως προαναφέρθηκε. Όταν μιλάμε για ένα έγγραφο στρατηγικής, περί εσωτερικής ασφαλείας, κυρίως στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, πρώτα απ' όλα αυτά πρέπει να οριστούν. Δεν είδα ορισμούς για την τρομοκρατία, για το οργανωμένο έγκλημα. Αναφέρεστε και στις μικροκλοπές παραβιάσεως πνευματικών δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι εκτός Εσωτερική ασφαλεία και τη σχετική στρατηγική. Είναι θέμα αστυνομική και δικαστική συνεργασίας. Πρέπει να επιληθούν στα πλαίσια άλλη στρατηγική. Πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν ανήκουν εδώ. Στη στρατηγική εσωτερική ασφαλείας. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα ήθελα πραγματικά να υπογραμμίσουμε ότι αν υπάρχουν συμπροματικά μέτρα για την εσωτερική ασφάλεια, για ριζοσπαστικά στοιχεία κλπ, θα πρέπει να υπάρχουν και ρήτρε διασφάλισης που θα περιέχονται στην στρατηγική. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί εκείνοι που είναι υπεύθυνοι τη ασφαλεία να προβλέπουν και να σπίζουν νέα μέτρα και να ακολουθούν οι υπεύθυνοι για θέματα δικαιοσύνη και να καθαρίζουν τα όσα έμειναν. Αυτό κάναμε τα τελευταία 10-15 χρόνια. Τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη προσέγγιση. Κάθε φορά που λαμβάνουμε νέα μέτρα, κάθε φορά που ακολουθούμε νέες στρατηγικές, θα πρέπει επίσης να φροντίζουμε για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα πρέπει να έχουμε και τις σχετικές ρήτρε ασφαλείας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Νομίζω ότι διατείνεστε ότι πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση της εφαρμογής. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρξαν υποθέσεις όπως μικρά εγκλήματα όπου το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως χρησιμοποιήθηκε και φαίνεται ότι είναι πολύ δυσανάλογο μέτρο. Σαν Επίτροπος, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε υποβάλλεται σχετική πρόταση να μετατρέψετε αυτό το μέτρο σε οδηγία που θα εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας θα είναι σημαντικό αυτό για μένα. Και μετά για τα ριζοσπαστικά στοιχεία που αναφέρατε, για τους εξτρεμιστές. Είναι κάτι που αναφέρατε και πριν. Καταλόγους με αυτά τα άτομα, οι βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα κρυφνή αυτά στοιχεία. Αυτό αφορά ορισμός. Τι είναι αυτό, τι είναι η ριζοσπαστική προσέγγιση αυτή, η ακρεφνής προσέγγιση. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί το πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε άλλου έξι στον κατάλογο, λέει ο πρόεδρο. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε σύντομοι για να μιλήσουν και οι άλλοι. Κύριε Μολτερ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομο. Η Κομισιόν μίλησε για τρομοκρατία και πόσο ξέρω υπάρχει και συντονιστής τρομοκρατίας στο Συμβούλιο. Για το ερώτημά μου είναι ποια είναι η συνεργασία μεταξύ ημών και του συντονιστή αυτού. Υποθέτω πως η απάντηση θα είναι εξαίρετη η συνεργασία. Αλλά το ερώτημα είναι, εάν αύριο έχουμε μια κρίση, ποιος είναι τελικά υπεύθυνο, είναι η Κομισιόν ή ο συντονιστής τρομοκρατίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Μπινκεβιτσιούτα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλστρομ για την παρουσίαση αυτής της σημαντικής, σημαντικότατης στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Θα πρέπει να γίνεται και συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και αρχών της Ευρωπαϊκή Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα και τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. Και όχι μόνο τα εθνικά κοινοβουλία, και οι πολίτες θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Γιατί, γιατί θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να αποφύγουμε τη στρατολόγηση πολιτών ε, σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Ένας άλλος ε, σημαντικός ε, παράγοντας είναι η οικονομική κρίση. Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε ε, εγκληματικά δίκτυα να εισέλθουν στον κρατικό μηχανισμό και σε κρατικούς φορείς. Επίσης πώς μπορούμε δηλαδή να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Τώρα, προστασία των εξωτερικών συνόρων. Σημαντική η προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για καταπολέμηση λαθρεμπορίου Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη επιθυμούν την προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη όπου οι τελωνιακοί υπάλληλοι τους τελευταίους δύο μήνες, Οκτώβριο και Νοέμβριο για παράδειγμα, δεν έχουν καν πληρωθεί. Γιατί τα κράτη-μέλη λόγω οικονομικής κρίσης ε, δεν έχουν χρήματα βρίσκονται σε εποχή λιτότητας κλπ. Οπότε πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι οι άνθρωποι που δεν πληρώνονται θα δουλεύουν σωστά. Θα ακούσω. Όλους ομιλητές τώρα γιατί δεν υπάρχει χρόνος για άλλο γύρο. κυρία Χάνκης. Κύριε Επίτροπε, να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή της τρομοκρατίας και πάντα λέμε πως πρέπει να αποφύγουμε παράλληλες δράσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για την εσωτερική ασφαλεία υπάρχει και μια εξωτερική πτυχή και αντιστρόφως. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την περιττή αλληλεπικάλυψη. Και να προσθέσω και μια τρίτη πτυχή. Πρόσφατα ακούσαμε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από ηγέτες του ΝΑΤΟ. Π.χ. Αναφέρθηκε πως το ΝΑΤΟ θεωρεί πως είναι όλο πιο σημαντικό να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Για να μην ε, γίνονται λοιπόν τα ίδια πράγματα παράλληλα. Πώς θεωρείτε πώς μπορούμε να κατανείμουμε τις αρμοδιότητες μεταξύ εσωτερικών, εξωτερικών αρχών και του ΝΑΤΟ, τους κάνει. των αρχών ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, τι, θεω τι άποψη έχετε για το ότι όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, τα κρατη ΜΑΕΛΗ ήταν υπεύθυνα για αυτήν. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αλλάξουμε αυτό και να γίνει κοινοτική αρμοδιότητα. Μια άλλη παρατήρηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, απάντησή σας γιατί σας είχα στείλει μια γραπτή ερώτηση για το ρόλο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της δημοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Νομίζω ε, πως αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι πολύ σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Εγώ το μεγαλύτερο μέρος ζωής μου το πέρασε μια κομμουνιστική χώρα και είχα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και τι βλέπω. Όλες αυτές οι ΜΚΟ παίζουν ένα σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται για ζητήματα κατασκοπίας. Όπως παραδείγματος χάρη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την απάντησή σας που αναφέρει δύο μελέτες ε, που συντάσσονται και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα ακούσουμε τα περιεχόμενα αυτών των μελετών γιατί θα είναι, είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Oui, merci. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο που ήρθε και την ευχαριστούμε για τις αφέστατες προτάσεις της. Εκτιμώ τη μέθοδο, έτσι δε περαιτέρω, διότι εδώ και καιρό οι τρομοκράτες έχουν θετήσει νέα στρατηγική, ολιστική, ολοκληρωμένη, που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οργανώνεται σε διεθνές επίπεδο. Άρα χαίρομαι ιδιαίτερος που η μέθοδος που προτείνεται να θετήσουμε είναι παγιωμένη, ενοποιημένη, που επιτρέπει να κατέξει αποτελέσματα. Πρέπει να είμαι σύντομη, αναφερθήκατε κυρία Επίτροπε, στην ύπαρξη περίπου 300 αποπειρών το χρόνο, ότι έλαβαν χώρα 300 απόπειρε ή τρομοκρατικέ απειλέ. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, διότι χρειαζόμαστε, κατά την άποψή μου, να έχουμε μια πολιτική που είναι πολύ σαφή εναντί των πολιτών μα, που ταυτόχρονα ανησυχούν οι πολίτε μα. Ανησυχεί όλη η Ευρώπη για την τρομοκρατική απειλή που είναι πάνω το κεφάλι μας και επίσης σωστά είναι πολύ που οι πολίτε όσον αφορά την χρήση, καμιά φορά χωρί προσοχή των προσωπικών στοιχείων ή μέτρα που λαμβάνονται και δεν κατανοούν πάντα αν έχουν η χρησιμότητα ή αν είναι καν αποτελεσματικέ. Αυτό που ζητείτε στα αεροδρόμια, π.χ. χάρη, όσον αφορά την χρήση των υγρών κλπ. Δεν ατηρείται αυτό παντού. Ε, αλλού εφαρμόζεται πολύ δραστικά και πιστεύουμε ότι από τις οδοντόκρεμες των εκατομμυρίων πολιτών περνά τα αεροδρόμια μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σοφά κατά πολλές τρομοκρατίες. Τώρα οι σαρωτές σώματος ε, είναι κάτι που αναφέρατε. Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι στον αφορά τις εγγύσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αφορά την χρήση των προσωπικών στοιχείων και την ελευθερία των ανθρώπων. Σε γι' αυτό. Και Ποιου κινδύνου θέλουμε να πολεμήσουμε στην ολοκληρωμένη αυτή μέθοδο που προτείνεται να θετήσουμε για να δράσουμε αλλά και για να προλάβουμε, τι θα κάνουμε για να εξηγήσουμε καλύτερα στου συμπολίτε μας που είναι εντό έλλειψη πληροφοριών. Όπως είδαμε με την υπόθεση Wikileaks που μας δείχνει ότι τα πάντα διατίθεται στο εμπόριο. Πώ θα μπορούμε να του προστατεύσουμε του πολίτε μα, για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αν είμαστε συγκεκριμένοι και ρεαλιστέ, νομίζω ότι θα είναι κάτι καλό. Παρακαλώ, συναδέλφοι, η Επίτροπο θα πρέπει να αποχωρήσει ένα λεπτό. Αν θέλετε να ακούσετε τι απαντήσει, να είστε σύντομοι. Άλλου δύο έχουμε στον κατάλογο. Η κυρία Ρομέρο Λόπε και ακολουθεί άλλη, αλλά έχει κλείσει το μικρόφωνο του Προέδρου και την ακούμε. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε, για την παρουσία σα. Ε, Σα έχω ξανακάνει την ίδια περίπου ερώτηση, θέλω να την επαναλάβω, σε ό,τι αφορά ε, τις μυστικών πληροφοριών των 27 κρατών μελών. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα, αλλά αν μιλάμε για μια στρατηγική εσωτερική ασφάλεια, ε, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη την δυνατότητα πρόληψη που έχουν οι υπηρεσίε μυστικών πληροφοριών ε, των κρατών μελών, αν κάνουμε κάτι τέτοιο, λέω, ε, είναι σαν να δημιουργούμε ένα κενό σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ αυτών των ε, υπηρεσιών μυστικών πληροφοριών. Μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών, για την ακρίβεια. Βέβαια, είναι πολύ πιο πολύ δυσχερή αυτή η συνεργασία, γιατί τα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν πω δεν θέλουν να ε, συντονίσουν ε, τέτοιου είδου πληροφορίε. Όμω δεν έχει νόημα οι μυστικέ υπηρεσίε πληροφοριών να κάνουν προσπάθειες ε, για την προάσπιση των εθνικών οικονομικών συμφερόντων της χώρας και να μην κάνουν το ίδιο για την ασφάλεια των πολιτών, είτε αυτής της χώρας είτε των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι καλύτερος συντονισμός, όχι μόνο ο συντονισμός σε συγκεκριμένες ε, ε, υποθέσεις, που έχει προταθεί. Ένας μηχανισμός συντονισμού πιο γενικός που θα έδινε τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ αυτών των ε, υπηρεσιών θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός από πολλά από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Γιατί, γιατί δεν υπάρχουν ε, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα ε, επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών και προσπαθούμε να είμαστε προληπτικοί. Πριν από λίγο καιρό, όταν είδαμε τις απόπειρε που έγιναν στι ΗΠΑ έγινε λόγο για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων των ΗΠΑ. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μηχανισμό ο οποίο ε, ε, θα επέτρεπε την συνεργασία, την αποτελεσματική συνεργασία, θα μα βοηθούσε πολύ. Για παράδειγμα, βλέπουμε τις, ε, το, το, site τη Wikileaks. Ε, χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία μεταξύ των ε, υπηρεσιών, ε, των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ε, διότι πολλές φορές παίρνουμε μέτρα τα οποία είναι δυσανάλογα. Οι, ζημιές που φυστάμε, φύστα την οικονομία, για παράδειγμα, είναι μεγάλες, αλλά χρειάζεται συντονισμό. Πολύ ωραία. Κύριε Ένστ. E. Ναι, έχω σου την παρενθετικά αυτό. Τρία πράγματα να αναφέρω. Πρώτον, θεωρώ πως τη στρατηγική αυτή, την οποία χαιρετίζω το ότι υπάρχει, ότι υπάρχει μια κοινωτική στρατηγική εδώ πέρα, πρέπει να ξανασκεφτούμε τη σχέση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Σε ποιο βαθμό όλα τα βήματα τα οποία έχουμε σκεφτεί εδώ πέρα ε, ανταποκρίνονται σκοπό και έχουν αναλογικότητα. πρέπει να το ξαναδούμε αυτό πριν μπούμε στις λεπτομέρειες. Δεν είναι δευτερεύον. Δεύτερον, αναμένω από εσάς ε, κυρία Μάλμστρομ να μας πείτε ξεκάθαρα τι είναι ριζοσπαστικοποίηση και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τρίτον, χρειάζεται οπωσδήποτε ε, να δούμε τι εννοούμε υπό την έννοια τρομοκρατία, υπό τις έννοιες αυτές. Εσείς μιλήσατε για τοπική τρομοκρατία, αλλά ε, υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών και σε σχέση με το τι εννοούμε στη ΣΥΠΑ. Πρέπει λοιπόν να το ξεχαρίσουμε αυτό και τελευταία παρατήρηση πάρα πολύ σύντομα ε, στο θέμα PNR. Συμφωνώ με την κυρία Σίπελ, πρέπει να δούμε τι κάνουμε πριν δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο και αν υπάρχει σκοπός να γίνει κάτι καινούργιο. χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεγάλη προσθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως μπορούμε να περάσουμε πολλές μέρες προσπαθώντας να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα να σκέφτεται κανείς το τι κάνει και να το αμφισβητεί. Αλλά εγώ δεν δέχομαι πω υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα. Ναι, μιλάμε για ασφάλεια. Ε, είναι θεμελιώδης δικαίωμα να μην ανατινάζεται κανείς, να μην ε, του κλέβουν τον τραπεζικό λογαριασμό ή την ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, επιτρέπονται όλα τα μέσα και όλες οι μέθοδοι. Όχι, πάντα υπάρχει αναλογικότητα, επικουρικότητα, προστασία των προσωπικών δεδομένων και το χρήσιμο κάθτος αναγκαίο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά είναι και η ασφάλεια δικαίωμα. Οπότε δεν αποδέχομαι πως κάτι δίνουμε και κάτι χάνουμε. Και η Κομισιόν και ειδικά εγώ προσωπικά σε στενή συνεργασία με την αντιπαράτατη την κυρία Ρέντινγκ πάντα προσπαθούμε να δούμε την πτυχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως υπάρχουν απειλές για τους ε, πολίτες και υπάρχουν βεβαίως πράγματι και βεβαίω μπορούμε να βγάλουμε μια μακροσκελή ανακοίνωση για την ίδια την ασφάλεια φιλοσοφικά βλέποντα το, αλλά πρέπει να δούμε αυτές τις τρει απειλέ και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και οι απειλέ υπάρχουν, Κάποιες είναι του οργανωμένου εγκλήματος, κάποιες ε, είναι απειλές από την φύση και πρέπει να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Τώρα, για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ναι, θα γίνει μια πρόταση, κυρία Σίπελ, για ευρωπαϊκά δεδομένα αεροπορικών επιβατών του χρόνου. Αυτό είναι στο πρόγραμμα της Οκόλμης, συζήτησαν ομόφωνα τα κράτη-μέλη. Σύντομα θα ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμαστε ένα εξωτερικό τέτοιο σύστημα και αν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο με τρίτες χώρες είναι θέμα του μέλλοντος, αλλά μιλάμε για ένα εσωτερικό τώρα πίεναρ. Και βεβαίως ευχαρίστω να συζητήσω την λογική, αλλά τα κριτήρια που έχουμε για τα εξωτερικά στοιχεία θα ισχύσουν οπωσδήποτε και ε, εσωτερικά για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ένταλμα σύλληψης. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ε, πώς θα αξιολογηθεί. Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Τα κράτη-μέλη βεβαίως ε, μπορούν πάντα να δουν ε, εάν υπάρχει κάποια κατάχρηση, εάν υπάρχουν ε, σαφή στοιχεία παραβίαση της οδηγίας ε, και του νόμου. Ναι κύριε Μίλντερ, πράγματι έχω στενή συνεργασία με τον κύριο Κέρκο, αυτός του Συμβουλίου για την Τρομοκρατία και πράγματι συνεργαστήκαμε στην σύνταξη αυτής της στρατηγικής. Βεβαίως δεν θα έχουμε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα σας ή στη χώρα μου αύριο. Εάν γίνει βεβαίως κάτι τέτοιο, ε, ο υπεύθυνο θα είναι ο ηγέτης της ε, κάθε χώρα. Βεβαίως μπορεί να απευθυνθούν στην Κομισιόν και να ζητήσουν βοήθεια, τεχνική βοήθεια, ιατρική βοήθεια, οτιδήποτε. Και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Αλλά στη τελική ανάλυση πάντα τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την ασφαλειά του. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμεί να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε τη συνεργασία, να δώσουμε μεθόδου, εργαλεία, οδηγίε, να ενισχύσουμε την κατεύθυνση που δίνουμε και να δούμε πώς μπορούμε να μοιράσουμε και να μοιραστούμε πληροφορίες. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο θέλουν τα κρατη αν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Λόπεζ, δεν θέλουν να μοιραστούν τις πληροφορίες τους τα κρατη με άλλες υπηρεσίες πληροφοριών. Το κάνουν ατύπως σε διμερή βάση, αλλά δεν παίρνουν τηλέφωνο και την Κομισιόν να μας πούνε τώρα θα δώσω αυτές τις πληροφορίες. Είναι λυπηρό αυτό, μας απογοητεύει καμιά φορά. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την ανταλλαγή κάποιων πληροφοριών που είναι σημαντικές για άλλα κράτη-μέλη, αλλά οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι εθνικές και εθνικές θα παραμείνουν. Κύριε Παγκεβούτση, θα γίνει μια πρόταση για την διαφθορά την ερχόμενη άνοιξη και αναμένουμε το ότι θα κάνει και η κυρία Μακοβέ εδώ πέρα. γιατί βεβαίως από εκεί διοχετεύονται τα λεφτά αυτά στον παράνομο τομέα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε θα δούμε πώς θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μηχανισμό, αλλά γίνονται ήδη αρκετά πράγματα στον τομέα της διαφθοράς. Και όπως είπατε δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο ε, μεγάλη αλληλεπικάλυψη και βεβαίως αντιλαμβάνομαι και αυτό που είπατε, πως, πώς να δουλέψουν τελωνιακοί άμα δεν έχουν πληρωθεί. Το βλέπουμε αυτό κατά περίπτωση και προσπαθούμε και να ενισχύσουμε και γενικά την ανάκαμψη της οικονομίας. Υπάρχει σταθερή σχέση βεβαίως μεταξύ, ξεκάθαρη σχέση μεταξύ εσωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας. Όπως θα θυμάστε ο κύριος Σολάνα παρουσίασε πριν από λίγα χρόνια μια στρατηγική εξωτερικής ασφάλειας ένα πολύ καλό έγγραφο. Εξακολουθεί να ισχύει γιατί η διεθνή συγκληματικότητα και η τρομοκρατία ε, κινείται και εκτός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε έχουμε συνεργαστεί εδώ πέρα πάρα πολύ με την Λέδη Άστον και τις υπηρεσίες της για να, προσπαθ... για να είμαστε όσο δυνατόν πιο έξυπνοι και να κινηθούμε στρατηγικά. Συμφωνώ Επίση κυρία Γκρίσμπεκ πω θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι στην επικοινωνία, πρέπει να έχουμε τα γεγονότα. Οι 300 απόπειρε που ανέφερα εγώ είναι τα στοιχεία τη Europol. Ε, δημόσια στοιχεία. Μπορείτε να βρείτε στατιστικά στοιχεία εκεί πέρα, αλλά και να δείτε το τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση. Και να καταβάλουμε μια κοινή προσπάθεια για να το μεταφέρουμε αυτό στους πολίτες, όχι να μην τους τρομάξουμε, απλά να ξέρουν το πρόβλημα. Νομίζω πως κάλυψα όλα. Βεβαίως ε, πολλές ερωτήσεις θα μας απασχολήσουν ξανά στο μέλλον και ευχαρίστω να έρθω στην επιτροπή σας. Και χαίρομαι και για την έκθεση η οποία θα μας δώσει μια ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα γιατί είναι δύσκολα και πολύπλοκα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσετε την ευκαιρία να έρθω στην επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμούμε το χρόνο που μας διαθέσατε και για να απαντήσετε. Σας ευχόμαστε καλή δουλειά. Ας πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Πάμε στο σημείο 14 και στο σημείο 15. Και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των συγγητών της κυρίας Μακοβέη, ζητώ συγγνώμη μάλλον από την κυρία Μακοβέη και από τον κύριο Έντσο για την καθυστέρηση. Συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βραζιλία για την απαλλαγή από την υποχρέωση τη τη βραχή διαμονή για του κατόχου κοινών διαβατηρίων και για του κατόχου διπλωματικών υπηρεσιακών ή επισήμων διαβατηρίων. Για το πρώτο θέμα η συγγήτρια είναι η κυρία Μακόβεϊ. Για το δεύτερο, η κυρία Ένση, 18 Απριλίου 2008 υιοθέτησε το Συμβούλιο απόφαση που δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει διαπραγματεύσει όσον αφορά τη ε, συμφωνία για την απαλλαγή από την υποχρέωση τη βραχία διαμονή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βραζιλία και τη τη διαπραγματεύσεων, τα δύο μέρη αποφάσισαν να συνάψουν δύο ξεχωριστέ συμφωνίε. Μία για τα κοινά διαβατήρια και μία για τα διπλωματικά υπηρεσιακά επίσημα διαβατήρια. Και επειδή συμφωνία για τα διπλωματικά υπηρεσιακά επίσημα διαβατήρια δεν χρειάζεται να επικυρωθεί από το Βραζιλιάνικο Κογκρέσο, μπορεί να προχωρήσει γρήγορα η επικύρωσή του. Καταρχά, θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει το περιεχόμενο των συμφωνιών και τις προτάσεις για απόφαση και μετά θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι ένας από τους ακρογωνίους λήθους της ε, πολιτικής θεωρήσεών μας είναι ο κανονισμός του 2001, πιο συγκεκριμένο 539 του 2001, που καθορίζει τη και το θετικό και το αντικό κατάλογο. Δηλαδή τον κατάλογο των χωρών που οι πολίτε του χρειάζονται θεωρείς όταν ε, ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο αντικό κατάλογος και ο, ο ε, θετικός κατάλογος είναι αυτέ οι χώρε των οποίων οι πολίτε δεν χρειάζονται. Ε, οι Βραζιλιάνοι πολίτες ε, βρίσκονται σε αυτό τον ε, θετικό κατάλογο, μπορούν να ταξιδεύουν στην ε, περιοχή Σέγγεν χωρίς θεώρηση. Μάλιστα πολλές χώρες έχουν και διμερείς συμφωνίες με την Βραζιλία για αμοιβαία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα κοινωνία κράτη-μέλη από την ημερομηνία ενταξή τους. Δηλαδή τα ε, κράτη-μέλη τα οποία εντάχθηκαν τελευταία έπρεπε να χορηγήσουν απαλλαγή θεώρηση στους Βραζιλιάνους πολίτες. Εκείνη την εποχή όμως η Βραζιλία δεν είχε διμερείς συμφωνίες με όλα αυτά τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερως με την Εστονία, τη Λετωνία, τη Μάλτα και την Κύπρο, οι οποίες ε, ε χώρες εξακολουθούσαν να, ε, να υποβάλλονται να υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρηση όταν ταξίδευαν στην ε, Βραζιλία οι πολίτες τους. Συνεπώ, ε, εξαιτία του μηχανισμού ε, αμοιβαιότητας έπρεπε και αυτέ να διατηρήσουν την ε, υποχρέωση θεώρηση. Η Κομισιόν ήρθε σε επαφή με την Βραζιλία, ήρθε σε επαφή με την Βραζιλία προκειμένου να καταργηθούν οι υποχρεώσεις αυτές. Πράγματι η Βραζιλία δεν είχε πολιτικούς λόγους να τις διατηρήσει, όμως εξαιτίας του συντάγματος ε, αυτή η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δεν μπορούσε να γίνει μονομερός, θα έπρεπε να γίνει ε, αμοιβαία μέσω μιας συμφωνίας. Από την άλλη μεριά τα τέσσερα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να διαπαραμετευθούν μετά την ένταξή τους τέτοιου είδους συμφωνίες με τη Βραζιλία, διότι το θέμα αυτό ε, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν ζήτησε εντολή να ε, προβεί στην σύναψη μιας ε, συμφωνίας απαλλαγής ε, θεώρησης με την Βραζιλία. Η εντολή αυτή δόθηκε το 2000, τον Απρίλιο του 2008 όπως γνωρίζετε και οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2009, αρχές του 2010. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο ήδη υιοθέτησε συμφωνία για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας η οποία έγινε στις αρχές του Νοέμβρη. Τώρα ε, θα ε, πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για την επικύρωση και το Βραζιλιανικό Κοινοβούλιο επίσης θα πρέπει ε, να δώσει τη συμφωνή γνώμη του με το κείμενο. Να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει μία μόνο συμφωνία απαλλαγής, αλλά δύο. Η μία αφορά τα διπλωματικά υπηρεσιακά και επίσημα διαβατήρια και μια δεύτερη συμφωνία για τους κατόχους κοινών διαβατήριων. Η Βραζιλία επέμεινε ιδιαίτερος ε, σε αυτό στη σύναψη δύο διαφορετικών συμφωνίων, διότι η διαδικασία επικύρωσης, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία είναι διαφορετική. Άλλη είναι για του κατόχου κοινών διαβατηρίων, ε, όπου το κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία, και άλλη για του κατόχου διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, για του οποίου η συμφωνία μπορεί να επικυρωθεί από την ίδια την κυβέρνηση χωρί να περάσει από το κοινοβούλιο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη ε, επικύρωση αυτή τη δεύτερη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δύο συμφωνιών, νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομο. Αυτή που αφορά του κατόχου διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων είναι πολύ απλή. Ε, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη συμφωνία για του κατόχου κοινών διαβατηρίων, πρέπει να σας, δώσω κάποιες, να σας πω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ε, η συμφωνία περιορίζεται σε άτομα που, εργα... που ταξιδεύουν για τουριστικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. 90 ως 95% του συνολικού αριθμού των ταξιδιωτών δηλαδή. Όμως η Βραζιλία επέμεινε να μην αφορά άλλες κατηγορίες οι οποίε προβλέπεται από την νομοθεσία του ότι δεν πρέπει να καλύπτονται από θεωρήσει μικρή διάρκεια. Καταρχήν, συμφωνήσαμε. Και το είχαμε ε, δεχθεί και σε ε, συμφωνίες με έξι μικρά ε, κράτη που είχαμε συνάψει νομονικές ε, πριν από μερικά χρόνια. Εκεί είχαμε εξαιρέσει για την ακρίβεια ε, ανθρώπους που ερχόντουσαν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χρειάζεται όμως να εξαιρέσουμε επίσης ερευνητές, φοιτητές, για μαθήματα κλπ. με την Βραζίλια. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνονται σε συμφωνίες απαλλαγής παλαιότερες ε, της δεκαετίας του 60 διμερός ε, συμφωνίες που είχαν συναυθεί διμερός με διάφορα κράτη-μέλη και τη Βραζιλία. Οπότε ε, θελήσαμε κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας με τη Βραζιλία οι πολίτες οι οποίοι δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα δυνάμει ε, παλαιότερων τέτοιων ημερών συμφωνιών να μην χάσουν τα προνομιά τους. Οπότε ε, η συμφωνία αυτή καλύπτει το τουριστικό και το επαγγελματικό ε, αλλά και επίσης προβλέπει ότι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες που προβλέπουν απαλλαγή συγκεκριμένων άλλων κατηγοριών εξακολουθούν να ισχύουν. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι δεν ακολουθούμε ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τέτοιου είδους διαφορές υπάρχουν ήδη και σε άλλα νομικά κείμενα. Για την Κομισιόν ήταν πολύ σημαντικό να εξασφαλίσει ότι η απαλλαγή θεώρησης ε, θα αφορά και τα τέσσερα ε, καινούρια ε, κράτη-μέλη τα οποία ανέφερα, με... γιατί και έτσι και αλλιώς με αυτή τη συμφωνία με τη Βραζιλία καλύπτουμε ε, τουλάχιστον 90% των ταξιδιωτών. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, λέει κύριε Μακοβέη. Ε, είναι δύο υποθ... Ε, ε, εντάσσονται στη διαδικασία συμφώνου γνώμη του Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζονται ουσιαστικέ τροπολογίε. Εγώ είμαι υπέρ του να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο για να συναυθούν αυτέ τι συμφωνίε ταχύτερο δυνατόν. Ούτω ώστε όλοι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όπω και εκείνοι Εστονία, Λετωνία, Μάλτα και Κύπρου, να ταξιδεύουν αν θεωρήσει του για τη Βραζιλία για τουρισμό και επιχειρήσει. Ε, το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα από τη γραμματεία τη ΛΥΜΠΕ είναι υποβολή ε, σχεδίων συστάσεων στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τέλος δηλαδή 31 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου, προθεσμία για τροπολογίες 11 ε, Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Μάρτιο 2011 και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο του 2011. Όμως θα ήθελα να ζητήσω από τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ να βρει πρώτερες ημερομηνίες για να το ταχύτερο δυνατόν. Δεν είναι επίμαχα θέματα, ε, δεν συζητούμε τροπολογίες, ε, πρέπει να επιβάλλουμε την αμοιβαιότητα στον αφορά τι θεωρήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, αμέσω. Αν ευκαθυστερήσουν, αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μόνικα. Ο κύριο Έντσιου έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λίγα πράγματα μπορώ να προσθέσω. Έχουν υποθεί τα περισσότερα. Όχι όσον αφορά τις δύο αλλά γιατί είναι απλά πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να μην ε, τις υποστηρίξουμε. Όμως, όπως είπε η κυρία Μακοβέη, πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία λίγο. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε μέχρι τον Απρίλιο, γιατί δεν νομίζω να είναι και κανείς κατά αυτών των οποίων προτείνονται εδώ πέρα. Έχω όμως μία παρατηρήση και μια που είμαστε εδώ πέρα σήμερα στην Επιτροπή μας και μιλάμε για απαλλαγή από θεωρήσεις, η παρατήρησή μου σχετίζεται με το εξής. Πάρα πολλές χώρες, ε, Ρουμανία, Τσεχία και Κύπρος ε, μεταξύ άλλων, δεν έχουν απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ε, για Ηνωμένε Πολιτείε και Καναδάς. Και Καναδά, ξέρετε πώς τα έχουμε συζητήσει αυτά τα πράγματα ξανά και ξανά και ε, έχω μια ιδέα την οποία θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω. Αλλά να δούμε τι μπορεί να γίνει με τις ε, χώρες αυτές. Ίσως η Κομισιό θα μπορούσε λοιπόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήπα ΕΕ Καναδά για τις απολαγές αποθεωρήσεων για άτομα τα οποία έχουν ε, υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια από τις χώρες αυτές ε, που δεν έχουν απαλλαγή. Αυτό κατά την άποψή μου θα ήταν ένα βήμα προόδου και σημαίνει πως ε, θα κάνουμε κάτι παραπάνω από το να κοιτάμε εκθέσεις. Έχουμε δει αρκετές τέτοιες φέτος μόνο φτάνει. Κύριε Μόλτερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπε ότι κατά 95% είχαμε ισότιμη κάλυψη όλων των πολιτών επαγγελμάτων και 5% είχαμε εξαιρέσει. Διότι για κάποιο λόγο η Βραζιλία επέμεινε επ' αυτού. Αυτή η αιμονή αφορά αποκλειστικά τη Βραζιλία ή ήθιστε στις περισσότερες συμφωνίες για θεωρήσεις που έχουμε διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε α, χώρα του κόσμου. Αφορά ιδιαίτερα τη Βραζιλία αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη έχουμε συνάψει έξι άλλες συμφωνίες εξαίρεση αποθεωρήσεις. Οι μόνοι που εχουμε διαπραγματευτει με οποιαδηποτε χωρα του κοσμου αφορα ιδιαιτερα τη από εκείνες τις συμφωνίες είναι εκείνοι που πάνε για κάποια δραστηριότητα που αμείβεται στον κανονισμό του 2001 που καταρτήσαμε θετικούς αρνητικού καταλόγου, τα κράτη-μέλη επέτρεπαν μονομερό την επιβολή θεώρηση για καναδού πολίτε Φερρυπίν, αν οι Καναδοί έρχονται για να εργαστούν. Ενώ Καναδάς, καταρχήν, οι Καναδοί δεν υποχρεούνται να έχουν θεώρηση για να ταξιδέψουν στο χώρο Σέγγεν. Αυτή η εξαίρεση υπάρχει στις υφιστάμενες ε, συμφωνίες. Οι άλλες εξαιρεσει στη συμφωνία με τη Βραζιλία αφορούν συγκεκριμένες χώρες. Ερευνητές που θέλουν να πραγματοποιήσουν έρευνες στα δάση, τα τροπικά, όπου θέλουν να προστατεύσουν τα δάση οι βραζιλιάνικες αρχές. Για διάφορους λόγους θέλουν να αφήσουν και άλλους, άλλες ομάδες από την εξαίρεση θεωρήσεως από τη συμφωνία αυτή. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε μελλοντικέ διαπραγματεύσει για συμφωνία δεν προτιθέμεθα να χορηγήσουμε τέτοιες εξαιρέσεις για άλλες ε, κατηγορίες. Ευχαριστώ. Σημειώσαμε δεόντως τα αιτήματα των δύο εισηγητών ή δυνατόν να ψηφίσουμε πιο νωρίς στην Επιτροπή τις εκθέσεις αυτούς, διότι δεν έχουμε τροπολογίες και μπορούμε να προωθήσουμε πιο γρήγορα τα χαρτοφυλάκια αυτά. Όπως γνωρίζετε, στο αρχικό πρόγραμμα της Επιτροπής μας προβλέπαμε συνάντηση συντονιστών από τις 11 μέχρι τις 12. Αυτό έγινε χτες όμως Οπότε μέχρι τις 12 έχουμε χρόνο και θα πρότεινα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και στις 12 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας για εγκληματικά για διάφορα εγκληματικά ζητήματα θα έχουμε τον Υπουργό Ντεκλέρκ της Βελικής Προεδρίας που θα μας κάνει μια παρουσίαση. Και ο Υπουργός θα έρθει μόνο στις 12 μας λέει η γραμματεία, αλλά πρέπει να περιμένουμε. για την Ευρωπαϊκή Έντολη Έρευνα σε ποινικέ υποθέσει. Σύντομο διάλειμμα. Α, κατέφτασε ο Υπουργό. Έχουμε τον εισηγητή όμως εδώ. Πέντε λεπτά διάλειμμα για να μαζέψουμε όλες τις δυνάμεις απαραίτητες.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 my colleagues, uh, συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη. Καθίστε παρακαλώ. So... Οπότε. Θα ήθελα να συνεχίσουμε το επόμενο σημείο. Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα σε ποινικέ υποθέσεις. Πρώτη παρουσίαση της πρωτοβουλίας 7 κρατών μελών για μια οδηγία για Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές προτάσεις στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, και μιλάει για την αμοιβαία αναγνώριση των περισσότερων μέρων μέτρων έρευνας με πολύ λίγους λόγους απόρριψης και έχουμε και πάλι την ευχαρίστηση να υποδεχόμαστε τον κύριο Ντεκλέρκα από τη Βελγική Προεδρία ο οποίος μας κάνει μια παρουσίαση της πρότασης αλλά πρώτα απ' όλα θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή τον κύριο Μέλο Ευχαριστώ Πρόεδρε θα κάνω την παρουσίασή μου στα πορτογαλικά, θα είμαι σύντομος. Χρησιμοποιώ την ε, γλώσσα μου όχι για λόγους αρχής, αλλά επειδή υπάρχουν πολύ τεχνικοί όροι, τους οποίους χειρίζομαι καλύτερα στην εθνική μου γλώσσα. Ε, έχει σχέση με την δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε θέματα ποινική φύσης. Όπως είπε η Πρόεδρος, είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και αφορά ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Εντάσσεται στο πλαίσιο δύο σημαντικών αποφάσεων, απόφαση πλαίσιο του 2003 που αφορά την, το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και μια άλλη απόφαση του 2004 σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή εντολή για ε, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικέ υποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο συντονισμός των κρατών μελών σε θέματα ποινικών ερευνών και ανακρίσεων. Όλα τα κρατημέλη επιθυμούν αυτές να γίνονται μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτή η πρόταση που εξετάζουμε ε, βασίζεται στην ε, παραδοχή ότι η συλλογή ε, αποδεικτικών στοιχείων είναι πολύ κατακαιρματισμένη και χρειάζεται ένα σύστημα συλλογής τέτοιων στοιχείων πιο αποτελεσματικό σε διεθνικό επίπεδο. Μία αρμόδια αρχή ζητά να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα έρευνα σε ένα άλλο κράτος μέλος. Και τα κράτη-μέλη τα οποία θα λαμβάνουν τέτοιου είδους ε, ευρωπαϊκές εντολές έρευνας θα πρέπει να την εκτελούν σύμφωνα με τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης. Βασικός ε, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να επιτρέψουμε ένα κράτος ε, μέλος, το εκδίδον κράτος μέλος, να εκδώσει μια ευρωπαϊκή εντολή έρευνας και να την κοινοποιήσει στο εκτελών κράτος μέλος, έτσι ώστε αυτό το τελευταίο να λάβει ένα ή περισσότερα μέτρα έρευνας για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Αυτή η ε, πρωτοβουλία είναι γενναία, θα έλεγα, ε, και χαρακτηρίζεται από ένα ευρωπαϊκό πνεύμα. Σίγουρα στο μέλλον θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της, των διαφορών των ποινικών συστημάτων ε, μεταξύ των ε, κρατών μελών, αλλά σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να βρίσκουμε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή και όχι αντίστροφα βέβαια. Θέλουμε ε, να μην γίνουν οι διαφορές αυτές σημαντικό πρόσκομα. Τελειώνω. Ε, αναφέροντάς σας το ιστορικό, η πρωτοβουλία ε, μάλλον διάφορα κράτη-μέλη ήδη έχουν καταθέσει τη θέση τους για αυτό το ζήτημα. Γερμανία, μέσω του Bundestag, ε, έγινε μια συνάντηση με όλα τα κόμματα. Το ίδιο έγινε και στην Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασία Δεδομένων επίση έχει υποβάλει την γνωμοδότησή τη για αυτή την πρόταση οδηγία στι 8 Νοεμβρίου. Στις 8 Νοεμβρίου ε, στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων ε, οι Υπουργοί Δικαιοσύνη ε, διεξήγαν μια πρώτη συζήτηση προ Ανατολισμού για το ίδιο θέμα. Μετά ζητήθηκε μια ανάλυση αντικτύπου από τον Γερμανό Υπουργό Δικαιοσύνης προς την Υπηρεσία Θεμελιών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επίσης ένας ε, βουλευτής της Επιτροπής ΑΛΔΕ, ο κ. Αλεξάνδερ, ο οποίος ε, ζήτησε μια, ε, επίσης μια ανάλυση αντικτύπου προς την ίδια υπηρεσία. Δεν ξέρω αν η διαδικασία που ακολούθησε ήταν σωστή, δεν πέρασε από τον εισηγητή, από τους κοιόδους εισηγητές, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, γνωρίζω ότι έχει αναλυθεί τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Δεν νομίζω ότι κανένας θα έχει αντίρρηση από όσο ξέρω, διότι δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε την ε, διαδικασία. Εγώ αυτό που πρότεινα είναι ε, να έχουμε μια προθεσμία, για παράδειγμα 15 Ιανουαρίου του 11 έτσι ώστε μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχουμε όλες τις απόψεις. Αυτή η πρόταση έχει λάβει όχι θα έλεγα επικρίσεις αλλά κάποιες ανησυχίες, κάποιους δισταγμούς που έχουν εκφραστεί εκ μέρους ορισμένων χωρών. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι δεν αναφέρονται τα θεμελιώδη δικαιώματα στι ποινικέ υποθέσει, για παράδειγμα το δικαίωμα τη σιωπή, ε, το δικαίωμα σε μια δίκαιη ακροματική διαδικασία κλπ. Ε, αναφέρονται μόνο δύο δικαιώματα, ε, όχι όμως και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, οπότε αυτό είναι ένα δισταγμός που έχει εκφραστεί. Η πρόταση αυτή αναφέρεται επίσης στις δικαστικές και μη δικαστικές αρχές ε, κρατών μελών. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει και τις αστυνομικές αρχές. Το Συμβούλιο στις 29 Οκτωβρίου είπε ότι εξαιτία τη νομική βάση δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι αστυνομικέ αρχέ. Αυτό είναι σημαντικό θέμα να το λάβουμε υπόψη. Ε, θα πρέπει, ε, λέει το Συμβούλιο, ε, η, στο εκδίδων κράτο μέλο, η αρχή που εκδίδει την απόφαση αυτή να είναι δικαστική και όχι μη δικαστική. Γιατί το αντίθετο θα μπορούσε να αντιβαίνει με την νομοθεσία και το Σύνταγμα πολλών κρατών μελών. Αυτά είναι ο απολογισμός της διαδικασίας μέχρι τώρα. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, σημαντικό. Περιμένουμε να εξελιχθεί θετικά. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ, κύριε Μέλο. Το εκτιμούμε, κύριε Λεκλέρκ, που, είμαστε, που είσαστε εδώ. Και θέλουμε και Ντεκλέρκ να μας παρουσιάσετε την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα, τα Ολλανδικά, επειδή είναι πράγματι ένα τεχνικό, τεχνικό θέμα, πρέπει νομίζω να είναι ξεκαθαρά τα πράγματα. Χαίρομαι λοιπόν κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Σιγητή, για το ότι ασχολούμαστε επί Βελγικής Προεδρίας ε, με αυτό το σημαντικό θέμα και δύσκολο, όπως είπε και ο εισηγητής. Είμαστε πράγματι πεπισμένοι πως ε, το νέο αυτό μέσο μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενισχύσει τις συνεργασίες ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν και τώρα δυνατότητες, ε, διάφοροι νόμοι, θέλουμε όλα αυτά να πάνε σε ένα ενιαίο μέσο. Οπότε είναι τεχνική η συζήτηση αλλά και επί της αρχής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης μας ε, και της συνεργασίας της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ε, στα νομικά συστήματα. Οπότε σας ευχαριστώ για το ότι εξετάζετε την Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνα ε, σε ποινικέ υποθέσει και είναι χαρά μου που σας την παρουσιάζω. Ε, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εστονία, Ισπανία, Αυστρία, Σλοβενία και Σουηδία κατέθεσαν αυτή την πρόταση από κοινού, οπότε έχει ήδη συζητηθεί αρκετές φορές ε, στο Συμβούλιο. Προσπαθήσαμε εμείς να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το γενικό πλαίσιο, καθώς και για κάποιες ουσιαστικέ πτυχές. Αλλά πράγματι θα είναι η Ουγγρική Προεδρία αυτή η οποία θα προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με σας. Τον Ιανουάριο δηλαδή. Το σκεπτικό είναι σαφές, είναι απλό. Θέλουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικέ υποθέσεις σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Σεβόμαστε δηλαδή ο ένας το σύστημα του άλλου. Ο στόχος αυτός ε, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, αυτό υιοθέτησε και το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου του 2009. Νομίζω είναι σαφές πως αυτό αποτελεί ένα λογικό βήμα στη διαδικασία υλοποίησης του ευρωπαϊκού χώρου ποινικών ε, θεμάτων. Θέλουμε λοιπόν απλοποιήσεις, θέλουμε να διευκολύνουμε το έργο των δικαστών, να σταματήσει ο κατακαιρματισμός, η σημερινή δηλαδή πρακτική. Θέλουμε ε, να σταματήσει, όπως είπα, αυτός ο κατακαιρματισμός όσον αφορά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχουν διάφορα μέσα, αποφάσεις πλαίσιο που θέλουμε να αντικατασταθούν από ένα και μοναδικό νομικό μέσο. Οπότε θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι εδώ πέρα μια ρήξη με το παρελθόν γιατί ήδη η σημερινή πρακτική υπάρχει. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ποιότητα. Να συνεχιστούν οι ορθές πρακτικές που έχουμε σήμερα, να ενσωματωθούν σε ένα νέο σύστημα επιπλέον. Βεβαίως θα δούμε και ποια είναι τα προβλήματα του σημερινού συστήματο και μιλάμε για απλοποιήσεις και επιταχύνσεις που θα επέλθουν και να απλοποιηθούν κάπως οι λόγοι απόρριψης, άρνησης, γιατί ένας από τους λόγους που μας οδηγεί αυτό είναι πως πάρα πολύ εύκολα κάποιες χώρες περισσότερο από άλλες απορρίπτουν τα αιτήματα συνεργασίας. Οπότε θέλουμε να απλοποιηθεί λίγο αυτή, αυτή η διαδικασία. Τώρα, οι στόχοι αυτοί δηλώνονται ε, από την δημιουργία του ευρωπαϊκού αυτού εντάλματος. Η ευρωπαϊκή αυτή εντολή έρευνας λοιπόν είναι μια δικαστική απόφαση η οποία απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος εκτέλεσης, να λάβει ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα έρευνας για να συλλέξει αποδεκτικά στοιχεία σε ποινικέ υποθέσει. Θα σα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Εάν παραδείγματο χάρη ένας Ισπανός είναι ύποπτος για α, δολοφονία και ε, ληστεία μεταφώνου σε βέλγικο έδαφος υπάρχει ένα αίτημα για να ερευνηθεί η κατοικία του στην Ισπανία. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποια σχέση επίσης με υπάρχον αποδεικτικό υλικό και αποδειχτεί πως θα πρέπει να υπάρξει μια περιγραφή λεπτομερής αυτού του υλικού θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας μόνο για την ανάκτηση των κλαπέντων υλικών ή άλλων συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων όπως π.χ. το, φόνο, το όπλο του φόνου. Οπότε η έκδοση Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας συν η έκδοση αιτήματος δικαστικής συνδρομής μπορεί να υπάρχει ή να έχουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα έρευνας, όπως π.χ. η έρευνα του σπιτιού κτλ. να ε, υπαχθούν στο αίτημα δικαστικής συνδρομής. Τώρα, η δικαστική συνδρομή που είναι μια γνωστή διαδικασία σημαίνει πως ο ανακριτής θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισμούς της Σύμβασης του 1995 για μεβαία αναγνώριση ποινικών υποθέσεων και τη Σύμβαση του 2000 για την ε, αμοιβή αναγνώριση ε, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής με τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν στην ε, συνθήκη αυτή. Οπότε, τι υπάρχει τώρα εδώ πέρα, κατακαιρματισμός και πάρα πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Οπότε, επιπλέον δεν προβλέπει δεν προβλέπουν τα μέχρι τώρα όργανα προθεσμίες, δεν προβλέπουν υποχρέωση επικοινωνίας Οπότε έχει ασχηθεί κριτική από πάρα πολλού δικαστέ και ανακριτέ οι οποίοι λένε Είναι σαν να πετάμε μπουκάλα στη θάλασσα αυτό το μέτρο. Δηλαδή δεν είναι σίγουρος κανείς εάν θα απαντηθεί σωστά η ερώτησή του και το αίτημά του. Υπάρχει μια ανασφάλεια η οποία έχει δημιουργηθεί από αυτά τα μέσα. Οπότε το Ευρωπαϊ... η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας θα δώσει τη δυνατότητα στο παράδειγμα που σας έδωσα στον Βέλγο ε, ανακριτή να λάβει όλα τα μέτρα έρευνας, ανάκριση, έρευνα κατοίκων, να μπουν όλα αυτά σε ένα έντυπο, να γίνει το αίτημα και να υπάρξει κάλυψη από ένα νομικό μέσο. Επιπλέον, η οδηγία αυτή και η συνεργασία με τις πανικές αρχές θα απλοποιηθεί θα επιταχυνθεί, θα υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των αρχών, δηλαδή δίνουμε βάρος πολύ στην επικοινωνία, συνεννοήσεις μπορούν να γίνουν με βάση κοινά μέσα για να γίνει και πιο σαφής και απλούστερη η επικοινωνία. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια ισορροπία και μεταξύ της νομικής ασφάλειας και της ευελιξίας. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ασφάλεια των πολιτών, να προστατεύσουμε και τα ατομικά δικαιώματα και πράγματι όπως λέει ο συγκητής είναι πολύπλοκο και καθόλου εύκολο το θέμα με το σημερινό κείμενο. Έχουμε διάφορες εγγυήσεις έτσι ώστε η θέση του υπόπτου και των υπολείπων εμπλεκομένων όπως των μαρτύρων να ε, οργανωθούν πολύ πιο απλά. Οπότε ε, η οδηγία παραπέμπει και αναφέρει συγκεκριμένα πως τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά επιπλέον. μια τέτοια ευρωπαϊκή εντολή έρευνας μπορεί να εκδοθεί μόνο σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Δηλαδή θεωρούν πως η δοκιμή αυτή από την αρχή έκδοση θα πρέπει να έχει γίνει. Επίσης, ο η δυνατότητα άρνησης ε, λόγω του ότι δεν είναι αξιόπινο κάτι άλλο σε μια άλλη χώρα δημιουργεί άμεσα προβλήματα καθώς θα πρέπει η αρχή η οποία θα εκτελεί ε, την εντολή αυτή να έχει την δυνατότητα να λάβει υπόψη τα ουσιαστικά στοιχεία, κάτι το οποίο βεβαίω ε, αντιβαίνει στην λογική τη αμοιβαία αναγνώριση όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη στο κράτος το οποίο εκτελεί να υπάρχει σεβασμός ως ε, κράτος το οποίο εκτελεί δεν μπορούμε απλά να το φέρνουμε σε δύσκολη θέση επιπλέον. Θα έχει πάντα η αρχή αυτή την δυνατότητα να ζητήσει και να κάνει άλλα μέτρα έρευνας από αυτά τα οποία ζητούνται στην περίπτωση στην οποία τα μέτρα έρευνας θα μπορούσαν να είναι λιγότερο καταναγκαστικά και να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αρνηθεί, αλλά μπορεί να πει πως εγώ σήμερα με την εθνική μου νομοθεσία μπορώ να ακολουθήσω εναλλακτικά μέτρα, τα οποία δεν θα είναι τόσο παρεμβατικά, αλλά οπωσδήποτε θα καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος χώρος ελιγμών. Επιπλέον η αρχή η οποία εκτελεί έχει αρκετές δυνατότητες να αρνηθεί. Υπάρχει ένας ε, λόγος όπως παραδείγματος χάρη το non bis in idem και άλλες τέτοιες γενικές αρχές ή για λόγους ε, ασυλίας. Υπάρχουν προνόμια. Υπάρχουν οι ουσιαστικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας όχι δημόσιας τάξης απλά, εθνικής ασφάλειας. Αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία μπορούν να στηρίξουν μια άρνηση εκτέλεση. Επίση λαμβάνεται υπόψη ε, ειδικά ο κατεπήγων χαρακτήρας ε, ορισμένων πραγμάτων, οπότε αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε για ένα καθεστώς το οποίο θα δίνει την δυνατότητα π.χ. άρνησης ενός τέτοιος αιτήματο ε, εντολής έρευνας εάν δεν υπάρχει κάτι το ανάλογο στη χώρα η οποία θα εκτελέσει την εντολή. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ανάλογη αξιόπινη πράξη μπορεί να το αρνηθεί. Επιπλέον προβλέπει η πρωτοβουλία συγκεκριμένους κανόνες για κάποιες ε, πολύ παρεμβατικές ε, ε, πολύ παρεμβατικά μέτρα έρευνα, όπω παραδείγματο χάρη υποκλοπέ, παρακολούθηση με βίντεο ή διαρκή σε πραγματικό χρόνο συλλογή στοιχείων, όλα αυτά ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω πω η εκτέλεση αυτών των μέτρων έρευνας τα οποία πρέπει πάντα να τα δούμε μπορούν να είναι και προς, ε, το, προς όφελος του υπόπτου. Ασάζ και αντισάζ, όπως λέμε. Οπότε, ακολουθούμε την αρχή, επίσης όσον αφορά το κόστος, ότι το κόστος το φέρει το κράτος το οποίο εκτελεί, αλλά συμφώνησε επίσης το Συμβούλιο πως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης, ότι δηλαδή ζητάμε πολυέξοδα μέτρα έρευνας και άρα δεν τα κάνουμε. Οπότε θα πρέπει να δούμε ε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν υπάρχει δυνατότητα να μοιραστεί το κόστος, κάτι για το οποίο βεβαίως είχαμε ευρύτατη στήριξη, οπότε προσπαθούμε να βρούμε το σύστημα αυτό, όπως σας είπα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να μπορούμε να μοιράσουμε το κόστος των μέτρων έρευνας. Γιατί βεβαίως θα πρέπει ε, να δούμε ε, αυτός ο οποίος ε, προκαλεί αν θέλει το έξοδο να το υπομειστεί κιόλας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο φάγκλος αυτός βρίσκεται σε μια πρώτη φάση, πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εντός του Συμβουλίου, αλλά η Βελγική Προεδρία το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην διαδικασία υλοποίησης του ευρωπαϊκού χώρου ποινικών, ποινικού δικαίου και είναι αυτό το οποίο θέλουμε είναι σταθερότητα και ποιότητα στο πώς θα αντιμετωπίζουμε τις ποινικέ υποθέσεις. Η Προεδρία λοιπόν την Παρασκευή θα υποβάλει μία έκθεση προόδου στο Συμβούλιο Υπουργών για να δούμε πού έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι συζητήσεις. Απλά κατ' ουσίαν δηλαδή λέμε το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και θα είναι η Ουγγρική Προεδρία αυτή η οποία μετά θα δώσει συνέχεια και ελπίζω με επικοδομητικό τρόπο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο και με το Κοινοβούλιο. Αλλά είναι κάτι το σημαντικό και κατά την άποψή μας ε, ουσιαστικό αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Ο λόγος του συναδέλφου, έχω πέντε μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο Κροτσέτα, Κίρκολτ, Άλμπρεκτ, Μάλτερ και Φόρς. Ο κ. Κορτσέτα. Κροτσέτα για την ακρίβεια. Αναφυσβήτητα το να φτάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνα είναι κάτι θετικό διότι επιτρέπει μια συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών δυνάμεων για να διώξουν με καλύτερο τρόπο, διώκουν καλύτερα το έγκλημα. Αυτή είναι μια απάντηση που φτάνει πολύ καθυστερημένα και παραλείπει διάφορα πράγματα από αυτά τα χρόνια η Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης θα έπρεπε να είχαν κάνει και αφορούν κάποιες υφιστάμενες δομές, αυτές που υπάρχουν ήδη εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως ενίσχυση της Europol, ενίσχυση του Eurojust, η έλλειψη παραξής του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα αυτής της φιγούρας, παρόλο που ζητήθηκε επανειλημμένα από το Κοινοβούλιο και συστήθηκε επίσης και από διάφορες δικαστικές αρχές εθνικές. Να υπενθυμίσω ότι ακόμα και ο δικαστής Φαλκόνε που δολοφονήθηκε μετά από τη μαφία ήδη είχε προτείνει τη δεκαετία του 80 να φτάσουμε σε τέτοια προσέγγιση. Σήμερα βλέπω να υπάρχουν λόγια στο κείμενο γίνεται αναφορά για αποτελεσματικότερη συνεργασία, ταχεία εφαρμογή κλπ. κλπ. Μία από τις λέξεις που αναλαμβάνεται συχνά είναι η ευελιξία, η έννοια της ευελιξίας. Πιστεύω ότι η ευελιξία είναι ο εχθρός του δικαίου. Διότι το δικαίο δεν βασίζεται στην ευελιξία, βασίζεται αντίθετα στην ακαμψία των νόμων και πάνω απ' όλα στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών. Όταν η έρευνα γίνεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για διάφορους πολίτες. Έχουμε κάποιες επικρίσεις όσον αφορά την πρόταση. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε αυτή την προσέγγιση. Εφόσον είναι διαθέσιμο το Συμβούλιο να το συζητήσει μέσω των εκθέσεων με το Κοινοβούλιο, ε, με τους κοιόδης ηγητές, είναι υπάρχει συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να, θέσω, δεν θέλω να θέσουμε εμπόδια, αλλά θέλουμε να θέσουμε διάφορα σημεία που θεωρούμε ότι είναι προβληματικά στην έκθεση. Το πρώτο ερώτημα. Στο κείμενο αναφέρεται γενικόλογα σε μία αρχή στην οποία θα κοινοποιείται το ένταλμα έρευνας. Μία αρχή γενική, αόριστη. Στη χώρα που εκτελεί το ένταλμα, κάθε χώρα μπορεί να καθορίσει. Να πει ότι η αρμόδιος είναι υπουργό Εσωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, κάποιος άλλος κάποιες φορές της κυβέρνησης. Κά... Κάτι που να μην συνάδει με το κράτος δικαίου ενδεχομένως. δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε εμείς όσον αφορά αυτή την ποικιλομορφία που απορρέει από την νομοθεσία στην Ευρώπη. Η χώρα μου γνώρισε το φασισμό και εμείς τρέμουμε στην ιδέα ότι μπορεί να διεξαχθεί από αστυνομικέ δυνάμεις αποκλειστικά η έρευνα χωρίς να υπάρχει καμία, κανένας έλεγχος από δικαστή. Εγώ πολλέ φορέ έχω απειληθεί από, τον, από τη μαφία και έχω καταδικαστεί και θάνατο από τη μαφία. Έχω κάθε συμφέρον λοιπόν να ενισχυθούν τα δικαστικά μέσα. Θέλω να γίνει αυτό, αλλά αυτό το μέσο μετά να μην ε, χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές, από τις πολιτικές δυνάμεις. Αναφέρεται το επίπεδο διαφθοράς που είναι διάφορη η διαφθορά στις αστυνομικέ δυνάμεις κάποιων χωρών. Σε κάποιες χώρες λένε ότι αν πάρεις μια κλίση στο δρόμο αρχίζει να, αρκεί να βάλεις να δώσεις κάποια χρήματα στον αστυνομικό για να διαγραφεί το πρόστιμο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο αστυνόμος ε, να κινείται χωρίς έλεγχο δικαστή, να πάρει το ένταλμα έρευνας. Ή κάποια αρχή παραλαμβάνει το ένταλμα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο αστυνόμος εκτελεί το ένταλμα χωρίς να περάσει μέσω δικαστού. Εγώ δημιουργούν τρόμο όλα αυτά. δεν γίνεται ο έλεγχος από πλευράς δικαστικών αρχών. Δεν ελέγχεται ε, η αστυνομία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Πιστεύω λοιπόν ότι οι αρχές δεν μπορεί να είναι έτσι αόριστα αναφερόμενες. Ποιος μπορεί να δώσει την έγκριση. Όχι μόνο τη διαδικασία α, συλλογής των αποδείξεων, που πρέπει να εγκρίνεται από δικαστή της χώρας που εκτελεί το ένταλμα. Δεν μπορεί γενικά να είναι κάποια αρχή κάποιος φορέας. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υποχρέωση να προωθούν, να εξελίσσουν την νομοθεσία των κρατών μελών, όχι να την κάνουν να υπαναχωρεί νομοθεσία των πιο φιλελεύθερων κρατών. Αντίθετα, πρέπει να βελτιώνουν την ομοθεσία των χωρών που δεν έχουν προχωρήσει τόσο. Από αυτή την έποψη μπορούμε να θεωρήσουμε ότι για ποινικά θέματα μπορεί να υπάρχει μια όριστη ε, ε, συνύπαρξη αμοιβαίας αναγνώρισης με διαφοροποιημένη προσέγγιση για την ίδια υπόθεση σε δύο-τρεις διαφορετικές χώρες να φεύγουν εντάλματα έρευνας. Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία. Και για μεμονωμένους πολίτες που αναφέρονται στην υπόθεση να υπάρχει διαφορετική ε, αντιμετώπιση αφορά την έρευνα και συλλογή στοιχείων με διαφορετικό τρόπο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και διαδικαστικά σε μια υπόθεση. Καταλήγω πιστεύω ότι θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες εναρμόνισης, ούτως ώστε το ένταλμα έρευνας και η μέθοδος που ακολουθείται και που συλλέγονται οι αποδείξεις δεν θα μπορεί να είναι διαφορετικές ε, και να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα έκδοση του εντάλματος και τη χώρα εκτέλεσης του εντάλματος. Με τους κρατούμενους προτείνεται η δυνατότητα μεταφοράς τους, ενδεχόμενη ανάκρισή τους, στη χώρα που εκδίδει το ένταλμα. Μετά υπάρχουν προβλήματα. Στην Ιταλία υπάρχει το 41α που είναι ειδικέ φυλακές για την κράτηση των μαφιόζων. Αυτοί κανονικά δεν μπορούν να έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Διότι ζήσαμε τραγωδία αυτά τα χρόνια με τη μαφία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν εχέγγυα όταν μεταφέρονται κρατούμενοι από χώρα σε χώρα, οι συνθήκες φυλάκισης δεν μπορεί να είναι ανώτερες ούτε κατώτερες. Θα πρέπει να είναι ίσες οι συνθήκες κράτησης με αυτές που έχει ο κρατούμενος στη χώρα στην οποία εκτεί την ποινή του, στη φυλακή. Συνάδελφοι, να είστε λογικοί ο ένας προς τον άλλο στην αντιμετώπιση σας, αλλιώς δεν μπορείτε να θέσετε και τις ερωτήσεις σας. Ο κ. Κίρκοπ είναι επόμενος που έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι συντομότερος. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα. Συμφωνούμε με την ιδέα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Έρευνας. Δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά ε, το, την διάρκεια ε, συνοδεύει το ένταλμα ε, σύλληψης είναι καλό να μπορεί να συλλέγει κανείς πληροφορίες με απλούστερο τρόπο με λιγότερη γραφειοκρατία. Όμως, και μιλώ όχι απλώς σαν συντονιστής, αλλά και σαν νομικός. Έχω κάποιες ανησυχίες. Ποιος είναι υπεύθυνο όσον αφορά την, το όλο εγχείρημα εδώ, αλλά και για τις πληροφορίες ανησυχώ. Ίσως να υπάρχει κάποια υποχρέωση. Δεν είναι θέμα συνεργασίας πλέον. Μιλάμε για υποχρέωση που επιβάλλεται από άλλη αστυνομική αρχή. Η παρόμοιο φορέα σε άλλη χώρα επιβάλλεται της Ευρώπης. Μπορεί να υποχρεώσει στη χώρα να ερευνήσει τη βάση δεδομένων DNA που διαθέτει. Σε κάποιες χώρες αυτό θα δημιουργούσε ανησυχίες. Μπορούμε σε διαφορετικές χώρες να ερευνούμε υποθέσεις που δεν αποτελούν εγκλήματα στη χώρα μας Υπάρχει και, ε, παραδείγματος χάρη, η εγκληματική κοφαντική δυσφήμιση στην Πορτογαλία. Θεωρείται έγκλημα, μπορεί να εκδοθεί ένταλμα στην Πορτογαλία, αλλά όχι αλλού. Υπό την παρούσα μορφή του εγγράμματο, η αδίποτε αστυνομική δύναμη θα μπορεί να ξεκινήσει έρευνα επί ξένου εδάφου όταν υπάρχουν ε, εύλογες υπόνοιες. Ποιος θα ε, διαφυλάξει τη σωστή εξέλιξη των διαδικασιών. Τι γίνεται με αποζημίωση νομική και διοικητική για οποιοδήποτε υποστεί βλάβες από αυτή την προσέγγιση που ακολουθείτε. Είναι πολιτική, πολιτικό θέμα πώς ζητά κανείς από τους πολίτες να το δεχτούν αυτό. Κάποιοι θα ανησυχούσαν πάρα πολύ γι' αυτό. Και πολλοί φορείς χρειάζονται όταν παραβιάζεται, παραδείγματος χάρη, ε, το άρθρο 8 ε, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τι γίνεται. Μιλώ υπό άλλη ιδιότητα τώρα. Σαν πρώην υπεύθυνο για θέματα πνευματικής υγείας, ψυχικής υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφέρθηκε και ο φασισμός πριν. Εγώ αναφέρομαι και στην Ανατολική Γερμανία. Οι αρχές τότε στην Ανατολική Γερμανία, τον παλιό κακό καιρό, ήταν χρησιμοποιούν πληροφορίες που αφορούσαν τα ιατρικά, το ιατρικό ιστορικό ή το ψυχιατρικό ιστορικό των πολιτών για να τους πιέσουν. Αυτά πρέπει να καλυφθούν, διότι μπορεί να έχουν αρχεία τέτοιου είδους οι αρχές. Και θα με ανησυχούσε τα μάλα αν οι ιατρικά στοιχεία, οι ψυχιατρικά στοιχεία διατίθοντος σε άλλη αρχή, σε άλλη χώρα, που αφορούσε οδήποτε πολίτη εκπροσωπώ εγώ στη δική μου χώρα. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, δεν θέλω να χρονοτριβήσω. Θέλετε να προχωρήσετε. Το κείμενο είναι αρκετά ατελές και εκείνοι που το προσυπόγραψαν στο κείμενο ίσως δεν το αντιλαμβάνονται καλά. Όλοι θεωρούν ότι είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν έκαναν τη δουλειά τους. Δεν είδαν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες αν εφαρμοστεί με κακό τρόπο. Όλοι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να σταματήσει η εγκληματικότητα και η πολύ μεγάλη εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα αλλά ο καλύτερο τρόπο να το πετύχουμε αυτό είναι να διατηρήσουμε την συνεργατική μα αυτή προσπάθεια και να προσθέσουμε περαιτέρω υποχρέωση για ορισμένα αρχή αν υπάρχει σωστό έλεγχο από την αρμόδια αρχή. Και από τη στιγμή που η ιδιωτική ζωή και τα θέματα προστασία των δεδομένων λαμβάνονται υπόψη. Εγώ θα το εξέταζα προσεκτικότατο το θέμα, όπω προχωράμε. Έχω κι άλλα να πω εν ευθέτω χρόνο, Αυτές είναι οι αρχικές μου παρατηρήσεις έχοντας ακούσει αυτά που άκουσα σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Κύρκο. Παρακαλώ συνάδελφοι να, να μιλήσετε μόνο για ένα λεπτό. Αλλιώς θα πρέπει να τελειώσουμε χωρίς να ακούσουμε τις απαντήσεις. Ο κύριος Άλμπρεχτ έχει το λόγο. Ναι, θα σύντομος, αλλά νομίζω πως οπωσδήποτε χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για την πρόταση αυτή. Ακόμα και αν συμφωνώ με τον κύριο Κέρκοπ πως ε, μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι απαραίτητη όσον αφορά την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων, αλλά θεωρώ πως είναι σημαντικό ακριβώς επειδή είναι σημαντική αυτή η πρόταση, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να την συζητήσουμε καλύτερα για το τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό και που χρειαζόμαστε κάποιες βελτιώσεις. Και εδώ πέρα οπωσδήποτε υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων, γι' αυτό χαίρομαι για τη συνεργασία με τον κύριο Μέλο και τους κύριους ηγητές. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, το θέμα της δημιουργίας κοινών αρχών. Για να δώσω άλλο ένα παράδειγμα μεταξύ των τόσων που δόθηκαν. Υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις συλλογής και αξιολόγησης αποδεικτικών στοιχείων. Π.χ. αν κάποιος ε, τον σταματήσουν στο δρόμο στη Γερμανία και το κάνουν αλκοτέστ και πρέπει να γίνει, να του πάρουν αίμα, μπορούν να τον εξαναγκάσουν στη Γερμανία. Στη Γαλλία δεν γίνεται αυτό, να πάρουν αναγκαστικά δείγμα αίματος γιατί πλέον δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Οπότε κάποιος ε, που βρίσκεται σε αυτή τη θέση είναι απλά ύποπτος. Και αυτό ε, βεβαίω είναι διανόητο στη Γερμανία. Οπότε είναι πολλά τέτοια παραδείγματα που έχουμε διαφορετικές διατάξεις για την προστασία ε, από την κατάχρηση και, και για την ε, απαγόρευση συλλογής στοιχείων και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε στις λεπτομέρειες και βεβαίως να αναπτυχθούν ε, με, την, ε, με βάση την ΕΣΔΑ και τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάποιες βασικές αρχές αλλά εγώ δεν θα ήθελα τώρα με την αμοιβαία αναγνώριση να πάμε τόσο πολύ χωρίς να έχουμε μία εναρμόνιση και χωρίς να εξετάσουμε λεπτομερώς ε, τις ε, διαφορές. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ οι προθεσμίες ε, για την εξέταση από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να μην είναι τόσο μικρές. Δεν είναι θέμα μερικών εβδομάδων, πρέπει να έχουμε απλά μια καλή πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μίλτερ. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Υπουργό. Έχω κάποια προσωρινά σχόλια. Ο Αλεξάνδρ Άλβαρο θα ήθελε να σας ανακοινώσει πως απίφθινε μια επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 126 του κανονισμού για να ζητήσει μια γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την πρόταση αυτή και ελπίζουμε πως σύντομα θα έχουμε αυτή την γνωμοδότηση. Πριν από τις 15 Ιανουαρίου δηλαδή του επομένου τους ε, βεβαίως οι συντονιστές νομίζω το συζήτησαν και το ενέκριναν. Ευχαριστώ κύριε Φως. Ευχαριστώ. Κάθε κράτος μέλος έχει ένα τελείως διαφορετικό σύστημα και διαφορετική νομική κουλτούρα, πολιτισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλιώς θα δημιουργηθεί μια νομική ανασφάλεια με ζητήματα τα οποία αφορούν πολύ θεμελιώδεις αρχές και θα έχουμε ένα ανοιχτό πεδίο για δημιουργία ανασφάλειας για πράγματα τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί. Γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πριν ε, δημιουργήσουμε τουλάχιστον καλύτερα, καλύτερες ελάχιστες προδιαγραφές για τους ε, υπόπτους και μετά να κάνουμε διασυνοριακές ε, συμφωνίες. Εντάξει, αυτή τη στιγμή λειτουργεί το σύστημα υπό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί. Εάν τώρα επέμβουμε από Ευρωπαϊκή Σκοπιά σε βασικές αρχές, τότε αυτό θα έχει φοβερές επιπτώσεις για το εθνικό σύστημα. Κατόπιν αναφέρθηκε πως ε, στη Γερμανία και πριν από την ε, Ανατολική Γερμανία είχαμε ένα άλλο σύστημα ε, που ήταν αυθαίρετο έναντι των πολιτών. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μπορούν να δρουν οι εκπρόσωποι του γερμανικού κράτους χωρίς νομική βάση. Επίσης μιλήστε για τους λόγους απόρριψης, άρνησης για το πώς μπορεί να αρνηθεί το κράτος εκτέλεσης. Εγώ έχω τελείω διαφορετική άποψη. Δεν μπορώ να αποδεχτώ η αστυνομική της δική μου χώρας χωρίς νομική βάση στο δικό μας το Σύνταγμα να δρουν. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνει μια εξέταση σύμφωνα με τις δικές του αρχές το κράτος εκτέλεσης. Υπάρχουν και άλλα σημεία, αλλά θα περιοριστώ σε αυτά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Κύριε Μέλλο, θέλετε να παρεμβείτε και με... σύντομα και μετά θα δώσω λόγο στον Υπουργό. Ναι, θα είμαι σύντομος. Να πω το εξή. Εγώ σημείωσα όλες τις παρεμβάσεις. Το θέμα είναι ευαίσθητο, το καταλαβαίνει ο υπουργό. Υπάρχουν αντιδράσεις. Ε, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανησυχίες ε, εθνικής φύσεως. Ε, εγώ είμαι δικηγόρος και έχω δουλέψει ως δικηγόρος και έχω δουλέψει πολλές εθνικές υποθέσεις και να πω συντονιστής ότι ο δικός μου σκοπός είναι να συναντηθώ όσο το δυνατόν περισσότερε φορέ με του σκιώδει ηγητέ, να συζητήσουμε λεπτομερώς για αυτό το θέμα, έτσι ώστε να βρούμε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Κάτι το, το οποίο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε κανένα κράτο μέλο. Για να μην ε, μπλοκάρουμε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Να πω τα εξή. Είναι σαφής μία συγκεκριμένη αντίρρηση. Αυτή αφορά τις ε, αρμόδιες αρχές ε, έκδοσης της έντολης. Ε, εμείς περιλαμβάνουμε και δικαστικές και μη δικαστικές αρχές. Εμένα δεν θα με πείραζε ένας δικαστής μιας χώρας με σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών να ζητήσει τη συλλογή ενό πιστηρίου σε μια άλλη χώρα. Το Συμβούλιο όμω λέει και μια αστυνομική αρχή, ένα αστυνομικό δηλαδή, να ζητήσει από δικαστή άλλη χώρας να συλλέξει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Στην Πορτογαλία, να σα δώσω ένα παράδειγμα, ορισμένα μέτρα πρέπει να υιοθετούνται και να επικυρώνονται από δικαστική αρχή, δεν μπορεί, από ανακριτή για παράδειγμα. Δεν μπορεί δηλαδή η αστυνομία ορισμένα μέτρα να τα εφαρμόσει χωρίς επικύρωση από το δικαστή. Κάποιο παρόμοιο, ένα παρόμοιο σύστημα εφαρμόζεται στη Γερμανία. Συνεπώς όλα αυτά θα πρέπει να τα σταθμίσουμε σωστά έτσι ώστε η πρωτοβουλία αυτή να μην αντιβαίνει με τα εθνικά συντάγματα. Θέλουμε όλοι αυτή η πρωτοβουλία να στεφθεί από επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό θα είναι προ όφελο όλων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Μέλου. Δίνω ξανά το λόγο στον Υπουργό. Θα ευχαριστήσω τους διερμηνείς να καταφέρουν και μείνουν μαζί μας μερικά λεπτά ακόμα. Um, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Είναι προφανές πως είναι ευαίσθητο το θέμα γιατί αγγίζει θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών μας. Και ε, πρέπει είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και έχουμε δύο βασικές κατευθύνσεις που μπορούμε να διαλέξουμε στην Ευρώπη. Την εναρμόνιση και να τα κάνουμε όλα ίδια. Και αυτό είναι και το δικό μου όνειρο. Και αρκετών. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε εδώ πέρα είναι πιο ρεαλιστικό. Δηλαδή κοιτάμε πώς μπορούμε να έχουμε αμοιβαίο σεβασμό των συστημάτων μέσω της καλύτερης συνεργασίας. Και να μπορέσουμε να εργαστούμε με βάση την αμοιβαία αναγνώριση, να έχουμε εμπιστοσύνη, σεβασμό για τα υπάρχοντα συστήματα. Όπου βεβαίως υπάρχουν όλες οι θεμελιώδεις αρχές. Οπότε ε, εκεί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, σε αυτό το σύστημα και πρέπει να προσέξουμε και εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτούς που λένε πως πρέπει να εναρμονίσουμε περισσότερα τα πράγματα και να τα κάνουμε πιο κοινοτικά. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό σε διάφορα σημεία. Προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε και το Letter of Rights την Παρασκευή. Αυτούς οι οποίοι ανακρίνονται ε, και να τους λέμε πως έχουν κάποια δικαιώματα τα οποία είναι ίδια για όλους και αυτό θα είναι πάρα, πολλά, πάρα πολύ θετικά είτε μιλάμε για μετάφραση, διερμηνήσεις κτλ. Να έχουμε μια εναρμονισμένη πρακτική θα γίνει και μία συζήτηση π.χ. για την παράσταση γόρου. για να τυποποιήσουμε και την ομολογία του δικαστηρίου. Αυτές είναι πολύ θετικές τάσεις εναρμόνισης. Τι κάνουμε τώρα. Βελτιώνουμε ένα υπάρχον μοντέλο συνεργασίας, μοντέλα με επιτροπές, ε, με διάφορες συνθήκες, αυτό το απλοποιούμε με σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Οπότε δεν είναι ότι κάνουμε ή το ένα ή το άλλο. Καμιά φορά κάνουμε εναρμόνιση, τώρα εδώ πέρα βασιζόμαστε στην αμοιβαία αναγνώριση. Πρώτον αυτών δεύτερον, συμφωνώ πλήρως να πούμε πως αυτό εδώ πέρα και το ε, είπαν πολλοί βουλευτές δεν ε, τίθεται ζήτημα, δεν γίνεται συζήτηση πως η εντολή έρευνας θα πρέπει να ε, επικυρωθεί αν θέλετε από έναν δικαστή ή κριτή. Δεν μπορεί μια αστυνομική υπηρεσία απευθείας να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη θα παίξουν ρόλο στον ορισμό ε, αυτού του πράγματος. Κάτι το οποίο θα είναι οπωσδήποτε με διαφάνεια. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανακριτή, θα, ε, όταν μιλάμε λοιπόν για δικαστική αρχή θα είναι ανακριτής, θα είναι δικαστής. Δεν είναι αυτά ταυτόσημα σε όλες τις χώρες. Θα πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει, μια δικαστική αρχή. Δεν θα είναι η αστυνομία που θα μπορεί να εκδίδει αυτές τις εντολές. και αντιστρόφως δεν θα τις εκτελεί. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική συνεργασία. Και αυτό λοιπόν συζητιέται ε, από τους υπουργού. Αυτό το οποίο δεν συζητάμε είναι η ε, λεγόμενη αυθαίρετη εντό οικών απόρριψη, άρνηση από μια χώρα η οποία λαμβάνει την εντολή. Πρέπει να έχουμε σεβασμό και προς το αίτημα. Οπότε θα πρέπει βεβαίω και αυτός που κάνει το αίτημα να σέβεται και να παίρνει σοβαρά την ε, αναλογικότητα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει όπως είπα δυνατότητα επαφής άμεσης. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα είδος να μην έχουμε μόνο μια αφηρημένη επαφή με έγγραφα μεταξύ των δικαστικών αρχών, γιατί οι δικαστές έχουν ούτως ή άλλως όλο και περισσότερες άμεσες επαφές και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία, αλλά δεν είναι δυνατόν η δικαστική αρχή του κράτους που εκτελεί να έχει μια αυτονομία και να κρίνει ε, μόνος του. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχουμε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες θα λέμε stop για λόγους θεμελιωδών ε, επιχειρημάτων. Ανέφερα παραδείγματο χάρη τις ε, ασυλίες, ε, των non bis in idem. Και πρέπει να δούμε πως θα πρέπει για εξαιρετικές, για πολύ βαριές περιπτώσεις να έχουμε ίσως περισσότερες δυνατότητες κάποια, δυνατότητες, κάποια εξαιρετικά μέτρα να μπορούμε να λάβουμε. Και αυτό θα είναι νομίζω απαραίτητο. Και θα προτείνω στο Συμβούλιο, στους Υπουργούς, να κάνουμε κάποιες διαφορετικές κατηγορίες μέτρων, ανάλογα με τη βαρύτητα των ε, μέτρων αυτών να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για τη χώρα η οποία εκτελεί να πει υπάρχει ένα πρόβλημα. Οπότε αυτή τη μέθοδο θα ακολουθήσουμε καθώς κάποιες χώρες ε, ήταν υπέρ αυτής της κατηγοροποίησης με απλούστερα και πιο πολύπλοκα μέτρα και ε, τις εξαιρέσεις όπως σας είπα. Οπωσδήποτε θα πρέπει κυρία Πρόεδρε, να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο ακόμα το θέμα. Είναι ευαίσθητο, με πολιτικές πτυχές οπωσδήποτε, αλλά υποθέτω πως ε, θα έχουμε και την απάντηση της υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι μια διαδικασία την οποία ε, συζήτησα με το Συμβούλιο Εντάξει, δεν πίστηκαν αμέσω, αλλά αν το ζήτησε το, το Κοινοβούλιο, το σεβόμαστε και ελπίζω πράγματι σύντομα να έχουμε μια απάντηση. Συμπερασματικά, ευχαρίστω είμαι στην ε, διάθεσή σας. Είναι ένα αναγκαίο εργαλείο, κάτι το οποίο ε, σημαίνει πως δεν έχουμε την ευελιξία να κάνουμε ό,τι θέλει το κράτος δικαίου εξακολουθεί να υπάρχει, απλά να έχουμε μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρώτη συζήτηση και ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους συζητητές για μια πιο θετική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Εντολή. Σας ευχαριστώ. Minister. Ευχαριστώ Υπουργέ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πρέπει να τερματίσουμε τη συνεδρίασή μας. Την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών θα διεξαχθεί σε 9 Δεκεμβρίου το απόγευμα από τις 3 το μεσημέρι και πέρα. Σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί, θα έχουμε ακρόαση